Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε τον κατάλογο των ομιλητών, βεβαίω, λέει η γραμματεία. So let's continue with the speaker. Ας συνεχίσουμε τον κατάλογο των ομιλητών από την προηγούμενη συζήτηση. Ο Σαμπάη από το Σλοβακικό Κοινοβούλιο έχει τον λόγο ως Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για το σχέδιο, αλλά έχω μερικές δεύτερες σκέψεις ε, για μερικές διατυπώσεις στο άρθρο 22 υπάρχει μια αναφορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αναλάβει ε, διπλωματικές προσπάθειες συμπεφωνημένες για να πείσει τους εταίρους στην περιοχή, όπως την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν, για την ανάγκη κοινή στρατηγικής απέναντι στην παγκόσμια πρόσκληση. Και διαρωτώ με, η Σαουδική Αραβία και το Ιράν έχουν, αν θέλετε, διαμέσου αντιπροσώπων ένα πόλεμο μεταξύ τους στη Συρία. Βασικά και το Ιράν. Δεν ξέρω. Έχω προβλήματα να ονομάσω το Ιράν εταίρο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, διότι το Ιράν επί δεκαετίες τώρα χρηματοδοτεί την τρομοκρατία, τρομοκρατικές ομάδες. Δημιούργησε την Χεσμολά, πρέμπτος χάρη, και πάνω από 50.000 ρουκέτες παρέδωσε στο Εσμπολά, εξοπλίζει και χρηματοδοτεί τη Χαμάς, πρέμπτος ε, χάρη. Δεν μπορούμε να ονομάσουμε λοιπόν τη χώρα αυτή μια εταίρο ε, για την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια ε, για να πάρουμε αυτές τις χώρες με τον πλευρό μας, αλλά έχω αμφιβολίες. Και στο άρθρο 25 υπάρχει μια φράση που αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας ως σημαντικό εταίρο στην επίλυση του κρίσης στη Συρία και στην καταπολέμηση κατά της ΔΑΕΣ. Νομίζω ότι και η Τουρκία επίσης είναι μέρος του προβλήματος και όχι εταίρο ε, για την επίλυση του προβλήματος. Η Τουρκία δεν καταπολεμάει την ΤΑΕΣ για την ώρα. Η Τουρκία βομβαρδίζει τους Κούρδους όπου αγωνίζονται κατά της ΤΑΕΣ. Αλλά και πάλι βλέπετε πόσο είναι δύσκολο να γράψει κανείς ένα κείμενο το οποίο να είναι ισορροπημένο και που να λαμβάνει υπόψη όλες ε, τις, όλες τις επιφυλάξεις, αλλά ήθελα απλώ να εκφράσω τις αμφιβολίες μου για ορισμένες ε, διατυπώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα πω τώρα σε λεπτομέρειες, ακόμα και αν είναι ενδιαφέρουσες μερικές από αυτές τις λεπτομέρειες. Όπως είπε και ο συνάδελφος από την Σεχική Δημοκρατία, εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για τα πρόσθετα βήματα τα οποία έχετε αναφέρει. Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο όμως έχει πραγματικά πάρει στα σοβαρά αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Από την αρχή λοιπόν, <clears throat> δηλαδή από την αρχή που είμαι Ευρωβουλευτή, το οποίο δεν είναι βέβαια μεγάλο χρονικό διάστημα σε σχέση με τη δική σα θητεία, είχα ζητήσει από την αρχή η Ευρώπη να δραστηριοποιηθεί, να πολύ πιο ενεργητικά για, τον, για τη σύγκρουση στη Συρία που έχει πολύ πιο άμεσες επιπτώσεις για την Ευρώπη από άλλες συγκρούσεις και ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι περισσότερο για την επίλυση αυτής της σύγκρουσης που φαίνεται δεν το έχει κάνει. Η Αμερική και η Ρωσία εμπλέκονται αυτή τη στιγμή στρατιωτικά. Εμείς <clears throat> με το ειδικό βάρος των 500 εκατομμυρίων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ίσως θα πρέπει και εμείς να ρίξουμε το βάρος μας για να μπορέσει να σταματήσει αυτή η αντιπαράθεση και πιστεύω ότι αυτά τα οποία είπε η κυρία Μογκερίνη σήμερα το πρωί ήταν θετικά και ελπίζω ότι αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε στο μέλλον μια πιο σημαντική δέσμευση στον τομέα αυτό στη Συρία. Υπάρχει όμως και ένας άλλος μεγάλος ελέφαντας στην αίθουσα, ο οποίος ίσως να ξεφούσκωσε λιγάκι τις τελευταίες 24 ώρες, αλλά εξακολουθεί να είναι μια μεγάλη απειλή. Πρόκειται για τον Ντόναλτ Τρόμπ. όταν και αν μίλησε για την ε, εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, αυτά που μας έλεγε ήταν λιγάκι ανατριχιαστικά. Και πάρα πολύ συγκεκριμένα, και εδώ επανερχόμαι στο ψήφισμά μας, θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτό που είπε ότι στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τα στρατέματα του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στην Ευρώπη, θα πρέπει η Ευρώπη να πληρώνει. και υπάρχει αυτή η συγκεκαλυμμένη απειλή από τη δική του πλευρά προς την κατεύθυνση αυτή. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν να δω κατά πόσο η πρόταση αυτή του Τραμπ αν κάπου συνάντησε κάποια μνήα, κάποια αντίδραση στο ψήφισμά μας και θα ήθελα λοιπόν, εάν όχι, να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιλανμόν, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομα. <clears throat> Μου φαίνεται θαυμασία η εκθεσή σας και πάρα πολύ πλήρε. Είναι μια πολύ καλή έκθεση. Εγώ έχω παρουσιάσει κάποιες σύντομε τροπολογίε, αλλά θέλω να τονίσω ότι την εκτιμώ πάρα πολύ θετικά. Θέλω να ε, επικροτήσω επίσης την έμφαση που δώσατε στην ανάγκη να δώσουμε μεγαλύτερη υποστήριξη στην πολιτική άμυνας και ε, ασφάλειας. Γιατί η ήπια δύναμη της Ευρώπης και μόνο δεν επαρκεί σε αυτές τις συγκυρίες. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό ότι και η κυρία Μογκερίνη υπεγράμμισε ακριβώς αυτό το σημείο. Ευχαριστώ πολύ. Λόπεθ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Αν μπορώ και εγώ να προσθέσω ορισμένα σχόλια στην έκθεση αυτή. Προφανώς έχει πολύ μεγάλη σημασία για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια πολύ δύσκολη πολιτική συγκυρία η πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Είναι απαραίτητο να ανταποκριθεί στι συγκεκριμένε συνθήκε που είναι πολύ διαφορετικέ από αυτέ που επικρατούσαν πριν από 15-20 χρόνια. Έχουμε τέσσερι ανοιχτού πολέμου στην περιοχή μα. Συρία, Ιράκ, Λιβύη, η Εμπένοι έχουν οδηγήσει σε αποτυχημένα κράτη <clears throat> στην γειτονιά μα. Βλέπουμε ότι γίνονται και πόλεμοι δύο αντιπροσώπων που εμπλέκουν τις μεγάλες περιφερειακές δυνάμεις όπως η Σαουδική Αραβία και το Ιράν. Έχουμε μια κρίση προσφύγων που δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά τη στιγμή που δεν έχουμε τον απαραίτητο θεσμικό σκελετό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε υψηλή τάσης εντάσεις οι οποίες γίνονται στο περιγύρο της Ευρώπης. Μέχρι πρόσφατα η πολιτική μας βασιζόταν στην ιδέα ότι το θετικό παράδειγμα Τη Ευρώπη θα οδηγούσε στο να ασπαστούν όλοι στη γειτονιά μα τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή ήταν τουλάχιστον η άποψη των ακαδημαϊκών μελετών για την περιοχή αυτή. Φυσικά αυτό δεν φάνηκε επαρκές. Πρέπει λοιπόν η διπλωματία μα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ασφάλεια και άμυνας, την ε, κατάλληλη πολιτική μετανάστευση και μια πιο ευφυή πολιτική για την ε, ανάπτυξη και τη συνεργασία. Και Όλα αυτά πρέπει να περιληφθούν στην πολιτική μας και φυσικά η πολιτική εξωτερικών θεμάτων θα πρέπει να συμπεριλάβει τα συμφέροντα που έχουμε, αλλά φυσικά θα πρέπει να εδράζεται και στι βασικέ αξίε και αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται να υπάρχει ισορροπία μεταξύ συμφερόντων και αξιών, <clears throat> όπω βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ώστε να έχουμε ένα πραγματικό εργαλείο για την ασφάλεια και την άμυνα τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο μικρόφωνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμένα θα με ενδιαφέρει περισσότερο να έχουμε μια απλοποίηση των δομών και μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών δομών στην Ευρώπη. Όταν υπάρχουν προβλήματα τα οποία δημιουργεί που δημιουργούνται, οι στρατιωτικοί θα πρέπει να ακούνε ποιες είναι οι πολιτικές απόψεις, αλλά και να μπορούν να εφαρμόσουν τις απαραίτητες ε, ενέργειες. Ο κίνδυνος είναι όλα αυτά που γίνονται για το στρατιωτικό τομέα να είναι απλώς χρήματα που πάνε στο βρόντο από την πλευρά των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ, λέγει και ο πρόεδρος. Τελευταίος, ο κ. Φανιούμπεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Αν εμείς σήμερα ανησυχούμε για το ενδεχόμενο τα επόμενα χρόνια οι Ηνωμένε Πολιτείε, ίσως όχι από τον Ιανουάριο, να μειώσει περαιτέρω την παρουσία της στην Ευρώπη, θα πρέπει ακόμα περισσότερο να σκεφτούμε για τη δική μας δέσμευση στην Ευρώπη. Πρέπει στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, στα πλαίσια της ε, συμμαχίας αυτής, να κάνουμε και περισσότερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των βαλτικών κρατών και ιδίω όταν τα βαλτικά κράτη ζητούν την έμπρακτη αλληλεγγύη μας. Και επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε και για την Ουκρανία. Η Ουκρανία μας ζήτησε μια αστυνομική αποστολή σε περιοχές που δεν γίνονται, ε, <clears throat> δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ακόμα μάχες. Πότε θα το κάνουμε αυτό. Εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε τα λόγια μας με πράξεις, τότε θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις χώρες οι οποίες θέλουν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Η Πολωνία, παραδείγματος χάρη, είναι μια από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκπληρεί το καθήκον του να έχει 2% του προπολογισμού της για την ε, άμυνα. Και παρόλα αυτά, για αυτό το λόγο, ορισμένοι την επικρίνουν. Αλλά δεν είδα να υπάρχουν οι αντίστοιχε κριτικές για χώρες και τις αρχές τους που επενδύουν πολύ λιγότερα στην άμυνα. Ευχαριστώ, Λέω για τη συζήτηση αυτή. Υπάρχει μια σειρά σημείων τα οποία θα λάβω υπόψη για την διατύπωση των ε, τροπολογιών συμβιβασμού που θα πρέπει να συζητήσω και με τους σκιώδεις εισηγητές. Κάποια από αυτά τα σημεία προέρχονται και από τα Εθνικά Κοινοβούλια, από τον Καρλ Σφάντσεμπεκ, σε σχέση με την ε, εξοπλιστική βιομηχανία. Ξέρουμε ότι υπάρχει και μία δυσπιστία μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας σε σχέση με τα θέματα αυτά της αμυντικής βιομηχανίας και γι' αυτό θα είναι δύσκολο να βρούμε έναν τρόπο να ξεπεράσουμε αυτό που είπατε. Αλλά και πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παροτρύνει τις χώρες να έχουν συνέργεια μεταξύ τους και ίσως θα ήταν χρήσιμο να έχουμε και μια μελέτη για τα αποτελέσματα μιας τέτοια ενδεχόμενη συνέργεια και της συνεργασίας των κρατών μελών στα θέματα αυτά, ώστε, όπως τον τα χρήματα των φορολογουμένων να χρησιμοποιούνται παράγοντας το κατάλληλο αποτέλεσμα που θέλουμε. Το ότι ένα άλλο ερώτημα που τέθηκε είναι ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα στη Συρία. Είναι απόλυτα σωστό αυτό, αλλά πώ. Όταν λέει κάποιο ότι πρέπει να είμαστε πιο ενεργοί εκεί, το ερώτημα είναι πώ. Είμαστε έτοιμοι να στείλουμε Γερμανού στρατιώτε, παραδείγματο χάρη, στην Συρία. Αυτό ελπίζω ότι δεν το λέει κανεί με αυτό το στόχο και αυτά που είπε ο Αυστριακός ε, συνάδελφος. Θέλετε να στείλετε τον Αυστριακό στρατό στη Συρία να πολεμήσει εκεί. Πρέπει να αντλήσει κανείς τα συμπεράσματα μιας τέτοιας ε, ε, δήλωσης. Υπάρχει θεωρητική ανάγκη να συμμετάσχουμε περισσότερο, αλλά οι συνέπειες είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια για να κάνουν πιο λειτουργική και επιχειριασιακή αυτή την αναγκαιότητα. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε και ποιες θα είναι οι συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας και θα πρέπει να το κάνουμε ό,τι χρειάζεται να κάνουμε ε, πιο συλλογικά. Και τώρα σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε. Δεν θα να κάνω τον Αμερικανό πρεσβευτή να περιμένει κι άλλο. Ich Σας παρακαλώ μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο πλέον. Έχουμε τώρα τον Αμερικανό Πρεσβευτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Γκάρνια. όποιος και αυτός με αδημονία περιμένει αυτή την ευκαιρία να δει τι θα προκύψει από τη σημερινή ημέρα, από τις εκλογές της ΗΠΑ και τη... και θα κάνει φυσικά ό,τι μπορεί για να μπορέσουν να παραμείνουν οι σχέσεις μας στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν θέλουμε να έχουμε άλλα σενάρια τρόμου. Ίσως θα πρέπει όμως να έχουμε και περισσότερη επίγνωση του περιεχομένου αυτών των ε, σχέσεων και ιδίως ε, σε ό,τι αφορά ορισμένα θέματα που έχουν να κάνουν με τις εμπορικές σχέσεις. Η Ευρώπη έχει μάθει ίσως κάποια διδάγματα από την ε, διαδικασία έγκρισης της Συμφωνίας ΣΕΤΑ και ίσως θα πρέπει να ανακατευθύνει λιγάκι την λειτουργία με έναν τρόπο που να οδηγεί σε αποτελέσματα και όχι μονάχα σε λαϊκιστικές κορώνες. Και εμείς θα πρέπει να δούμε αυτό το θέμα των εμπορικών σχέσεων με μια συνολική άποψη που λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα μιας τέτοιας συμφωνίας για όλους μας. Η περίπτωση της ΕΤΑ ήταν ένα αρνητικό παράδειγμα του πώς <clears throat> δεν πρέπει να συνάπτουμε συμφωνίες όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη εμπορική δύναμη. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο την ε, συμφωνία αυτή και να βασιζόμαστε μονάχα στα εθνικά ή τα υποεθνικά συμφέροντα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Έχετε το λόγο εξοχότατε. Well, no predictions about tonight. Δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις σήμερα το βράδυ καταρχάς. Αλλά με βάση την έκβαση των σημερινών εκλογών ενδεχομένω δεν είναι και η τελευταία μου παρέμβαση σε αυτή την Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω κάνοντας κάποιες παρατηρήσεις προσωπικής φύσεως. Καταρχάς, ως πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα έλεγα ότι το αξίωμα αυτό ήταν μια δουλειά, ήταν μια πραγματική αποστολή, ένα λειτουργήμα, ένα πραγματικό πάθος. Ξυπνάω κάθε πρωί και πιστεύω πραγματικά στο έργο μου. Θυμάμαι όταν είπα στον 13χρονο γιο μου το 2013 ότι με είχαν διορίσει πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με κοίταξε μορθάνικα τα μάτια και σχεδόν δεν με πίστευε. Και μου είπε εσύ, εσύ θα αναλάβεις αυτό το αξίωμα. Και πραγματικά αυτό ανήψε στο ηθικό μου μπορώ να πω. Και το θυμάμαι αυτό, το θυμόμουν πολλέ εβδομάδε και μήνε μετά και προσπαθούσα πραγματικά να ανταποκριθώ κι εγώ στο ερώτημα αυτό. Γιατί εγώ και όχι κάποιο άλλο. Πιστεύω γιατί καταρχά πιστεύω στην Ευρώπη, πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μητέρα μου ήταν Ιταλίδα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι κατά το ίμιση Ιταλό. Η γυναίκα μου είναι Ισπανίδα. Τα παιδιά μου ζουν και μεγαλώνουν στο Λονδίνο και αισθάνονται ότι είναι εξίσου Ευρωπαϊο όσο και Αμερικάνοι. Και τα τελευταία χρόνια τη ζωή μου, όπω γνωρίζετε, τα έχω περάσει στην Ευρώπη. Πιστεύω κράτοντα λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 25 χρόνια και για ποιο λόγο πάλι εγώ, γιατί πιστεύω πραγματικά στις, ε, στην ισχύ της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών και το κοινό καλό. Και δεν είναι διπλωματικά λόγια αυτό το οποίο λέω, δεν είναι μια διπλωματική ρητορική, είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνω και βιώνουμε θεωρώ κάθε μέρα. Πιστεύω πραγματικά και στο δικό σας το θεσμικό όργανο ότι εσεί συμβάλλετε πάρα πολύ στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και θεωρούσα ανέκαθεν ότι οι στενές σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποτελούν ένα αναπόσπαστο τμήμα της θητείας μου. Έχω έρθει σε επαφή με όλες τις πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία δυόμιση χρόνια και τον επόμενο μήνα θα είναι το επόμενο και τελευταίο έβδομο ταξίδι που θα κάνω στο Στρασβούργο και θα χαρώ πάρα πολύ πραγματικά να δω για άλλη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πλήρη λειτουργία στο Στρασβούργο. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που μπορώ να απευθυνθώ σήμερα σε εσά. Καθότι λαμβάνουν χώρα βέβαια οι προεδρικέ εκλογέ σήμερα το βράδυ. Έλμαρ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, σε ευχαριστώ για τη φιλία σου. Και Ελάχιστοι πολιτικοί στην Ευρώπη γνωρίζουν τόσο καλά τις Ηνωμένε όσο εσύ και ελάχιστοι πραγματικά έχουν τόσους φίλους και από τις δύο πλευρές. Σαφώς πρέπει να μιλήσουμε και για τα αποτελέσματα των σημερινών εκλογών, καθότι υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει τόσο η Ευρώπη όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η στάση της Ρωσίας, η προκλήση της Ρωσίας, η προσφυγική κρίση, η ανώτια γειτονία της Ευρώπης που ζητά μια συντονισμένη διατλαντική προσέγγιση. Οι Ηνωμένε Πολιτείες θα χρειαστούν μια ενωμένη ισχυρή Ευρώπη ανεξάρτητα με το ποιος θα αναλάβει τελικά το προεδρικό αξίωμα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Αντενάουρο είχε πει ότι η Ευρωπαϊκή Ενότητα ήταν το όνειρο λίγων και έγινε η ελπίδα πολλών σήμερα και αποτελεί αναγκαιότητα για όλους μας. Το όνειρο αυτό εξακολουθεί και παραμένει ζωντανό παρά όλες αυτές τις προκλήσεις και κάθε μέρα θυμάμαι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν πολύ σημαντικούς εταίρους σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από πάρα πολλή αναστάτωση. Μετά το Brexit έλαβα πάρα πολλά τηλεφωνήματα και ήρθα σε επαφέ με πάρα πολλούς αρμοδίους. Πάρα πολλοί μου λέγανε ότι θα πρέπει να εμφυσίσω νέα εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά αναρωτιόμουν και εγώ για ποιο λόγο δεν υπήρχαν περισσότεροι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ευρωπαϊκό και το εθνικό επίπεδο που θα μπορούσαν πραγματικά και αυτοί να αντιταχθούν στα καταστροφικά σενάρια τα οποία είχαν αρχίσει να παρουσιάζονται εκείνη την εποχή. Είναι στρατηγική σημασία αυτό, δεν είναι απλώς μια πολιτική marketing, μια πολιτική ενημέρωση και επικοινωνιακή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι πολίτε να μπορούν να βλέπουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα συγκεκριμένο όραμα, ότι μπορεί και αντιμετωπίσει σημαντικέ προκλήσει όπω προσφυγική κρίση ή η τρομοκρατια Ο Υπουργό Εξωτερικών Κέρι, όντω, όταν είχε έρθει στι Βρυξέλλε, μίλησε για τα ζητήματα αυτά. Ο πρόεδρο Ομπάμα επίση στο Ανόβερο τον Απρίλιο του 2016. Αν η Ευρώπη παραμείνει μεμονωμένη, δεν θα καταφέρει σε καμία περίπτωση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες μιας παγκοσ... ενός κόσμου ή τις ευκαιρίες του ελευθέρου παγκοσμιμένου εμπορίου και ουσιαστικά δεν θα είναι αντάξιος εταίρος της ε, Αμερικής. Αν χάσει την εμπιστοσύνη της στο μέλλον της, αν χάσει την εμπιστοσύνη της στις αξίες της, τότε θα γίνει όλο και πιο ευάλωτη σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά θέλουν να βάλουν κατά του ε, δημοκρατικού, οικονομικού, ανοιχτού μοντέλου, το οποίο πρεσβεύουμε. Ουδέποτε το ευρωπαϊκό εγχείρημα δεν ήταν τόσο ψηλά στις προτεραιότητες των ΗΠΑ. Μολονότι πρόσφατα είχαμε μια απόφαση από το Σταγματικό Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, θεωρώ ότι το Brexit είναι πιο πιθανό τελικά να συμβεί από τον αποτραπή. Προφανώς σεβόμαστε τις αποφάσεις των Βρετανών πολιτών, και βέβαια η απόφαση αυτή επηρεάζει πολλές αποφάσεις όπως για παράδειγμα η κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η πολιτική κατά των κλιματικών αλλαγών, η πολιτική για την ενέργεια και πραγματικά ανησυχούμε για το αν θα καταφέρουμε να κρατήσουμε την ισορροπία μεταξύ ήπιας και πιο σκληρής δύναμης. Παραμένω όμως αισιόδοξο. Δεν θεωρώ ότι μόνο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε και ο Ζαμονέ, δυναμώνεται περισσότερο μέσα από τις κρίσεις, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να λάβουμε συλλογική δράση. Η διαδικασία διαπραγματεύσεων για το Brexit θα πρέπει να είναι όσο δυνατόν πιο γρήγορη, δίκαιη, αμερόληπτη και ελπίζω ότι ε, η μελλοντική σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι όσο το δυνατόν πιο επικοδομητική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το Brexit να μην συμβεί με άτακτο τρόπο, γιατί αυτό θα είναι ιδιαίτερα επιζήμιο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την Αμερική. Στα πλαίσια τη διατλαντική αυτή κοινότητα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την επιθετική αυτή Ρωσία. Η Ρωσία προχωρά σε όλο και πιο προκλητικέ ε, δράσει. Ε, έχει δεχθεί πάρα πολλέ καταγγελίε από μη κυβερνητικέ οργανώσει, καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα, δολοφονεί πολλέ φορέ του ε, αντιπάλου τη και προσπαθεί να αναταράξει τελικά τις βασικές αρχές δομές πάνω στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το Κέντρο Στρατηγικών Διεθνών ε, Σπουδών έχει δημοσιεύσει το έγγραφο αυτό που λέγεται The Kremlin Playbook, πώς μπορούμε να κατανοήσουμε πραγματικά την επιρροή της Ρωσίας στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με τα ζητήματα αυτά τα επόμενα τέσσερα χρόνια όλοι μας. Η πρώτη γραμμή του πυρός βέβαια εξακολουθεί και είναι η Ουκρανία, όπου ε, Προσπαθούν βέβαια οι άνθρωποι εκεί να αποτρέψουν την, τις επεκτατικές τάσεις της Ρωσίας, είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε μέσω της Ουκρανίας να αντιμετωπίσουμε το κλεπτοκρατικό μοντέλο του Πούτιν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να συνεχιστούν οι προσπάθειες και πραγματικά χαιρετίζω την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ουκρανία, προκειμένου να αρχίσει να εξακολουθεί να ασκεί πίεση στη Ρωσία αν καταρρεύσει η Ουκρανία, ουσιαστικά αποτυχάνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα καταφέρουμε ουσιαστικά να καταφέρουμε να προασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εδαφική ακαιρεότητα. Και αν δεν μπορούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσουμε και να προασπίσουμε τι βασικέ αυτέ αρχέ, εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ θα καταφέρουμε να το πράξουμε εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αρκεστούμε σε ημίμετρα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να επιβάλλουμε κυρώσει κατά τη Ρωσία μέχρι να αρχίσουν να εφαρμόζονται οι αρχέ της συμφωνίας του Μίνσκ. Και πρέπει επίσης να δούμε και ποια είναι η στάση της Ρωσίας απέναντι στα Δυτικά Βαλκάνια και στις χώρες της ανατολικής γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ρωσία πολλές φορές προσπαθεί να παρεμποδίσει τον δρόμο των χωρών αυτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς το ΝΑΤΟ. Γίνεται μια καμπάνια παραπληροφόρησης από τη Ρωσία η οποία προσπαθεί να επηρεάσει και την όλη συζήτηση πολιτικής που γίνεται. Εμείς υποστηρίζουμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και όλους αυτούς τους οργανισμούς οι οποίοι μάχονται για την ανεξάρτητη πορεία αυτών των κρατών. Επίσης, είμαστε κατά του αγωγού Nord Stream 2 μεταξύ ε, Ρωσίας και Γερμανίας μέσω της Βαλτικής. Ουσιαστικά αυτό θα παρακάμψει την Ουκρανία και κατά αυτόν τον τρόπο θα στερήσει τη χώρα αυτή από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε τέλη διαμετακόμισης. Ουσιαστικά ο αγωγός αυτός ε, δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση ούτε τις χώρες προέλευσης ούτε τις χώρες προορισμού και είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί μια απόφαση το συντομότερο δυνατό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίζω ότι εσεί θα συνεχίσετε να ασκείτε πίεση. Ήδη έχετε καταβάλει πολύ σημαντικέ προσπάθειε. Η πρόσφατη απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανοίξει την πρόσβαση προ τον αγωγό πάλι ουσιαστικά δεν είναι θετικό νέο, γιατί θα αυξήσει το ρόλο πάλι τη Ρωσία. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση και είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαφοροποιηθούν οι δρόμοι ενεργειακής παροχής ενεργειακού εφοδιασμού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει επίσης να καταφέρουμε να συμβάλλουμε στην ειρήνευση στη Συρία. Έχουμε ένα τεράστιο πεδίο μάχης, το οποίο έχει οδηγήσει σε πάρα πολλές καταστροφές και πάρα πολλούς θανάτους, ένα τεράστιο αριθμό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ανακοίνωσαν την απόφασή τους να αναστείλουν τις διμερείς συζητήσεις με την Ρωσία όσον αφορά την, ε, ε, την ανακοχή, καθότι η απόφαση αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη. Δεν έχουμε καταλήψει προφανώ του πολίτε τη Συρία και προφανώ επιδιώκουμε την ειρήνη στην περιοχή. Θα κάνουμε κάθε το δυνατό μέσω τη Διεθνή Ομάδα Υποστήριξη τη Συρία, μέσω των ΗΠΑ και άλλων οργανισμών, προκειμένου να καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Κάνουμε προσπάθειε προκειμένου να απαλύνουμε τον πόνο των Σύριων πολιτών και ε, μέσω της στρατιωτικής και της διπλωματικής οδού προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους 67 παγκόσμιους εταίρους μας στην περιοχή. Πρέπει να μειώσουμε επίση τον αριθμό των ανθρώπων αυτών που αναγκάζουν να καταλήψουν τα σπίτια του. Και καταλαβαίνετε ότι οι προσφυγικέ αυτέ ροέ δημιουργούν τεράστια προβλήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητήματα εθνική ταυτότητα, ζητήματα αλληλεγγύη, ζητήματα σχέσεων με τα Δυτικά Βαλκάνια και με την Τουρκία Ζητάμε λοιπόν από τους ε, Ευρωπαίους ηγέτες να αντιμετωπίσουν με ανθρωπιστικό και ανθρώπινο τρόπο τις μεταναστευτικές αυτές ροές. Και πάλι το δικό σας το Κοινοβούλιο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για το ζήτημα αυτό και ουσιαστικά έχει ζητήσει μια ευρωπαϊκή λύση στην προσφυγική αυτή κρίση. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες μας πρόσφατα είχε να κάνει με την υπογραφή Τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Συνέβαλε πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε και καταφέραμε τον τελευταίο αυτό διάστημα πριν από μερικέ μέρε να θέσουμε επίσημα σε ισχύ τη συμφωνία αυτή. Θα χρειαστεί όμω μια διατλαντική συνεργασία και ηγετική θέση προκειμένου να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία. Τέλο, όσον αφορά το TTIP, παραμένουμε δεσμευμένοι στι διαπραγματεύσει προκειμένου να έχουμε μια φιλόδοξη συμφωνία TTIP. Ακόμα και αν το είπατε και αυτό εσεί κύριε Πρόεδρε, ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή ασχολείται με κάποια πολύ θεμελιώδη ζητήματα. Πώ θα καταφέρει δηλαδή να εξισορροπήσει την συμμετοχή των κρατών μελών και πώ θα καταφέρει να κάνει τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν με ισορροπημένο τρόπο σε μια πολύπλοκη τελικά συμφωνία. Ελπίζω θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια οριστική λύση. Αν δω λίγο την εντολή μου, αν δω λίγο τη θητεία μου, θεωρώ ότι έχουμε σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έχουμε δημιουργήσει τον απαραίτητο αυτό μηχανισμό προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των αρμόδιων αρχών πάλι όμως έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Ο πρόεδρος Ομπάμα κατέστης, δημιούργησε μια αμερικανική πλέον νομοθεσία το Φεβρουάριο του 2016 προκειμένου να υπάρχει μια νομοθεσία πλέον που θα επεκτείνει τα δικαιώματα των Αμερικανικών των Αμερικανών πολιτών και που να μπορούν να καλύπτονται και οι Ευρωπαίοι πολίτες από την κάλυψη αυτή που προπαρέχεται στις ΗΠΑ. και θα έχετε τη δυνατότητα να προσυπογράψετε και στη συμφωνία αυτή στο άμεσο χρονικό διάστημα και ελπίζω θα το κάνετε. Η διατλαντική εταιρική σχέση είναι πάρα πολύ σημαντική και μόνο αυτή μπορεί να διασφαλίσει την παγκόσμια σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία. Και αυτό δεν έχει συμβεί μόνο τα τελευταία 70 χρόνια, αλλά θα διασφαλίσει την ισορροπία αυτή και την ασφάλεια και για τα επόμενα χρόνια. Η καταπολέμηση της δημαγωγίας του λαϊκισμού θα αποτελέσει μια καθοριστική πρόκληση την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω τις ερωτήσεις σας και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε και μια ουσιαστική συζήτηση. Our TLD, uh, από την αντιπροσωπεία του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ο κ. Μόντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας εκθέσω μια παρατήρηση και δύο ερωτήσεις. Εγώ καταρχήν θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι απόλυτα τις τελευταίες σας Διατυπώσει Είναι απαραίτητη η συνεργασία σε στρατηγικό επίπεδο με τις ΗΠΑ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω ότι αυτά που θα γίνουν απόψε το βράδυ στις ΗΠΑ δεν θα αλλάξουν την στάση των ΗΠΑ επί τη βάση των κοινών αρχών και αξιών και βάσει της κοινή μας ιστορίας. Τα ερωτήματα. Εγώ έχω, είμαι σίγουρος ότι έχετε παρακολουθήσει αυτά που έγιναν εδώ στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την έγκριση της συμφωνίας ΣΕΤΑ. <clears throat> την ε, σημασία που είχε αυτή η διαδικασία για την Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα για τη Βαλονία, για ένα μηχανισμό επίλυση των διαφορών, το οποίο, ο οποίο μηχανισμό θα ισχύσει και στην TTIP. Θα ήθελα να σα ε, ρωτήσω πώ βλέπετε το μέλλον τη TTIP μετά από αυτά που έλαβαν χώρα με την ε, ΣΕΤΑ. Το δεύτερο μου ερώτημα, ίσω το έχετε απαντήσει ήδη, το μέλλον των σχέσεων μα με τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι σημαντικός παίκτη σε παγκόσμιο επίπεδο, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μια ενεργειακή και στρατιωτική δύναμη, <clears throat> παρά όλα αυτά που έχουν γίνει με τις παραβιάσεις του, του, διεθνούς δικαίου, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση του προβλήματος της τρομοκρατίας, για την επίλυση της Συρίας, ακόμα και αν έχει μια λαθασμένη στάση. Πώς βλέπετε λοιπόν το, το μέλλον των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, Αμερικής και Ρωσίας μετά από την θητεία της κυρίας Κλίντον ως Υπουργού Εξωτερικών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Πρέβζη. Ήταν ε, πάρα πολύ έντιμη η παρουσίαση εισαγωγή όταν αναφέρατε τις προκλήσεις ε, που μας περιμένουν ε, την καταπολέμηση της δημαγωγίας και του λαϊκισμού. Ελπίζω απόψε το βράδυ ότι θα κερδίσετε όσον αφορά σε αυτή την πρόκληση όταν θα έχουμε το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών. Ερώτηση. Μερικοί λένε όταν, όταν πρόκειται για εξωτερική πολιτική δεν έχει σημασία ποιος θα κερδίσει από τους δύο υποψήφιους. Μπορείτε να να μας πείτε εσείς ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές, τι θα διαφέρει όσον αφορά την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που που ε, και εσείς λέτε ότι είστε Αμερικανοευρωπαίος και ότι βεβαίως αντιλαμβάνεστε τα πράγματα με πολύ έντιμο τρόπο, με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντική ημέρα αυτή για όλους. Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα σε αυτό που με εξέπληξε περισσότερο στην προεκλογική εκστρατεία για τις διατλαντικές σχέσεις, τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έγινε λόγος ως προς το μέλλον των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Έχετε μια εξήγηση, αναφερθήκατε στην συμφωνία TTIP. Υπογράψαμε τη ΣΕΤΑ με μερικές δυσκολίες. Ποια είναι η θεώρησή σας των πραγμάτων σε σχέση με το θέμα αυτό. Έχετε δει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη διαχειρίστηκε τις διαπραγματεύσεις για τη ΣΕΤΑ. Τελευταίο σημείο σήμερα το πρωί συζητήσαμε λεπτομερώς με την Φεντερικά Μογκερίνη σε σχέση με την παγκόσμια στρατηγική όπου συνηγορεί υπέρ μιας συνεργασίας πιο ολοκληρωμένης ανάμεσα στις ε, δυνάμεις, στις μεγάλες δυνάμεις. Ξέρετε ότι έχουμε καλές σχέσεις, θέλουμε να τις διατηρήσουμε, αλλά θέλουμε επίσης να θεσπίσουμε μια ευρωπαϊκή άμυνα. Όχι απλώς περισσότερη συνεργασία, αλλά περισσότερη συνεργασία, ολοκληρωμένα μέσα, ε, περισσότερο προϋπολογισμό, περισσότερο συνασπισμό. Ποια είναι η θέση σας σχετικά με τα θέματα της ευρωπαϊκής άμυνας. χωρίς ε, μικρόφωνο. Κύριος Χατζηγεωργίου. Νομίζω ότι έχετε την καλύτερη παρουσία ε, σε αυτήν ε, την Επιτροπή και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό που είπε το παιδί σας και στη θέση την οποία υιοθέτησε. Μιλήσατε πολύ για το λαϊκισμό και θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα λέχθηκαν. Ο κύριος Στάμπ έχει ε, λαϊκισμό σε όλα τα στοιχεία των ομιλιών του ο κύριος Τραμπ. Και αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα, να δω μια τέτοια χώρα να έχει τόσο λαϊκισμό στις ομιλίες του ενός εκ των δύο υποψηφίων. Αυτό σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν υπάρχει εκπαίδευση σε αυτή τη χώρα υπάρχει το να σκεφτεί κανείς ότι ο κύριος Τραμπ θα μπορούσε εύκολα να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είπατε ότι η συνεργασία ανάμεσα στις Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ζωτική σημασία. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, δεν βλέπετε ότι εμείς ε, ε, δηλαδή ε, το Ηνωμένο Βασίλειο εκπροσωπεί όταν εκπροσωπείται από τον Τόνι Μπλερ, ότι εσείς και αυτός ήταν ε, στο πρόβλημα στην Μέση Ανατολή όταν με τον κύριο Μπλερ πήγαμε στο Ιράκ, τώρα έχουμε 500.000 ανθρώπους που πέθαναν. Τι σκέφτεστε για το θέμα αυτό. Μπορούμε να ξανασκεφτούμε, να αναθεωρήσουμε την εξωτερική μας πολιτική. Και τέλος θα ήθελα να σας ρωτήσω, βλέπετε καμία πρόοδο στις συζητήσεις για να λυθεί το πρόβλημα της Κύπρου. Παρακολουθείτε το θέμα αυτό, το πρόβλημα αυτό, διότι τώρα υπάρχει κάποια κινητικότητα και υπάρχει ε, στο, στην Ελβετία υπάρχουν ε, συνομιλίες. Δεν θα... Βεβαίω δεν θα ήθελα να ξανασκεφτείτε την έκπληξη που σας προκάλεσε το παιδί σας. Αν <coughs> βλέπω ότι όλοι έχουν ε, γίνει υποψήφοι για καγκελάριο στη Γερμανία, πρωθυπουργοί στην Ελλάδα. Δεν θα ήθελα να κάνω σχόλια για τα συστήματα παιδεία των δύο χωρών, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ για την ε, ε εισαγωγή σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Γιατί είπατε ότι η Ουκρανία είναι τόσο σημαντική για την ασφάλειά μας και την αυτονομία μας στην Ευρώπη, κάτι το οποίο το κατανοώ βέβαια, αλλά στην περίπτωση αυτή, γιατί έχουμε εμπάργο όπλων, γιατί αφήνουμε την ε, Ουκρανία να είναι μόνη της με ένα εξοπλισμό ο οποίος είναι ανεπαρκές ενάντια της στρατιωτικής μηχανής της ε, Ρωσίας. Δεύτερο ερώτημα σε σχέση με την TTIP. Εγώ θεωρώ ότι είναι αποφασιστική για τη διατλαντική σχέση. Σας δίνω δίκιο <clears throat> σε ό,τι αφορά τα εμπορικά θέματα και τις εμπορικές σχέσεις. Γιατί όμως θα πρέπει αυτή η συνθήκη να μπει τόσο βαθιά στο νομικό μας σύστημα και τις δημοκρατικές μας δομές. Εγώ νομίζω τα δύο πράγματα θα πρέπει να μείνουν χωριστά. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Εξοχότατε. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για την ειλικρίνειά σας. <coughs> Τουλάχιστον τα πράγματα γίνονται σαφή. Καταλαβαίνω ότι και ο πρόεδρος μου, ο κ. Μπρόκ, είναι ένας ε, υπηρέτης των ΗΠΑ. Νόμιζα στην αρχή ότι υπηρετούσε την Ευρώπη, αλλά βλέπω ότι πιο πολύ προτιμά τις ΗΠΑ. Δεν πρέπει να σας... Ε, δεν σας καταπραίνω σε σχέση με την ρωσική προπαγάνδα. Όχι, δεν έχει αποτέλεσμα εδώ. Τη δική σας προπαγάνδα ακολουθεί το Κοινοβούλιο και όχι τη ρωσική προπαγάνδα και δεν έχει χώρο η ρωσική προπαγάνδα εδώ και στη συνέχεια θα ήθελα να σας θέσω ορισμένα ερωτήματα σε σχέση με την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η Ρωσία είναι επιθετική δύναμη, είπατε. Στο Ιράκ είναι η Ρωσία επιθετική δύναμη. Στο Ιράκ και τη Λιβύη ήταν η Ρωσία ο επιτιθέμενος. Ή μήπω ήταν οι Ηνωμένε Πολιτείε που παραβίασαν το διεθνές δίκαιο παρεμβαίνοντας. Το ίδιο για την Ουκρανία. Υπάρχει περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη διαφάνεια, λιγότερη ε, διαφθορά από ό,τι στο παρελθόν στην Ουκρανία. Περισσότερη ανάπτυξη. Όχι. Και σας λέω, λέτε για την ρωσική προπαγάνδα, μα δεν υπάρχει σε αυτό το κοινοβούλιο και δεν υπάρχει στην Ευρώπη και στους μεγάλους θεσμούς που δικούν την Ευρώπη. Τέλος για το λαϊκισμό. Ο λαϊκισμός είναι η φωνή των λαών που υποφέρουν. Η πραγματικότητα πάντα αναδύεται στην πολιτική και θα το δείτε και στη χώρα σας γιατί και ο Τραμπ είναι ένα φαινόμενο που έχει να κάνει με την κοινωνιολογική και οικονομική κατάσταση ενός λαού που υποφέρει. Δεν μπορείτε να βγάλετε από την, πραγματικότητα, από την εικόνα την πραγματικότητα αυτών που υποστήριζουν τον Τραμπ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρεσβευτά. Ευχαριστώ. Βλέπετε ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας, λέει ο κύριος ε, Μπροκ. Ο κύριος Τάνοκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε κύριε Γκάρνερ. Εγώ ελπίζω θα παραμείνετε ως πρεσβευτής για κάποιο διάστημα στο μέλλον, όχι μονάχα γιατί ήσασταν εξαιρετικό στο ρόλο αυτό, αλλά και γιατί είσαστε φίλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για όλους μας το να είναι ο Τραμπ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, να έχουμε κάποιον ο οποίος είναι φίλος του Πούτιν και να, υπο... και να ηγείται του ελεύθερου κόλπου. Εγώ αναρωτιέμαι πώς κάποιος ως, όπως ο Τραμπ έχει φτάσει τόσο κοντά στα ηνία της εξουσίας. Φαίνεται ότι ζούμε σε μια πολιτική κατάσταση που δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Εγώ αγωνίστηκα για να αποτραπεί το Brexit και συμμερίζομαι τη λύπη σας για το γεγονός ότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Ελπίζω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα βοηθήσουν την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και το λαό του Ηνωμένου Βασιλείου να μείνουν κοντά στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι ο ρόλος σας είναι πάρα πολύ σημαντικός και ένας μεγάλος ατλαντιστής όπως ο Λάμ Φόξ του Ηνωμένου Βασιλείου δεν πιστεύει ότι το να αποσυνδέσουμε το Λονδίνο από την τεσσερακονταετή και σύνδεσή του με την Ευρώπη δεν, ότι δεν πιστεύει ότι θα βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα γίνει για το αν υπήρχε μια προεδρία Κλίντον τον Ιανουάριο. Θα είναι πιο στεναρή στον παγκόσμιο στίβο σε ό,τι αφορά την δυνατότητα παρέμβασης από τον πρόεδρο <clears throat> Ομπάμα, ο οποίος ήταν πολύ καλός πρόεδρος, αλλά μετά την ε, εμπειρία του Αφγανιστάν και του Ιράκ ήταν πολύ επιφυλακτικός για να παρέμβει. Και έχασε ίσω μια ευκαιρία στην Συρία, γιατί βλέπουμε τώρα τι τεράστιε και τρομερέ σφαγέ που γίνονται στο Χαλέπι από τι ρωσικέ βόμβε. Αναρωτιέμαι αν η πρόεδρο Κλίντον θα είναι υπέρ μια μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλεία για να αποτρέψει στο μέλλον να γίνονται αυτά τα εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα, τον βομβαρδισμό των εφοδιοπομπών του Ηνωμένων Εθνών που γίνεται δυνατή λόγω της ε, αδράνειας και αβελτηρίας των δομών του, του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πιστεύω λοιπόν ότι με τη Χίλαρη Κλίντον θα μπορούσαμε ίσως να μπορέσει η Δύση να αποτρέψει την άνοδο αυταρχικών χαρακτήρων, ε, καθεστώτων μάλλον, στην Κίνα ή στη Ρωσία που θα οδηγήσουν ίσως σε μελλοντικές ομότητες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Κόουσο. Χαίρομαι για την παρουσία σας. Όπως είπε ο κύριος ε, Μπροκ, η δημοκρατία έχει και το μεγαλείο της. Αλλά εμένα μου φαίνονται αυτά τα οποία λέτε, μου φαίνονται λυπηρά, γιατί ο λόγος σας ήταν ψυχροπολεμικός, ήταν επιθετικός. Μιλάτε για μια επιθετική Ρωσία. Αλλά τι πρέπει να πει κανείς για τις ΗΠΑ με τόσες στρατιωτικές βάσεις σε όλο τον κόσμο. Με μια τεράστια ε, στρατιωτική δύναμη. Μιλάμε για την, αν συγκρίνουμε τώρα την παρεμβατικότητα της Ρωσίας και τη δική σας, θα θυμηθείτε ότι στη Λατινική Αμερική έχετε μια μεγάλη ιστορία παρέμβασης και έχετε ευθύνη για πάρα πολλά πραξικοπήματα στη Λατινική Αμερική, παραπληροφόρηση. Μία περίπτωση που τη γνωρίζετε πολύ καλά, το Ιράκ. Είπατε ψέματα. Μα εμπλέξατε σε ένα τρομερό πόλεμο. Γιατί στο, στην περίπτωση του Ιράκ φτάσατε ακόμα και στην δολοφονία δημοσιογράφων. Στη Λιβύη επίσης. Θα ήθελα να ξέρω τι έχει γίνει τον 1,5 χρόνο Τη μεγάλη συμμαχία εναντίον του Ισλαμικού κράτου. Ούτε ένα εκατοστό εδάφου δεν έχει επιτευχθεί. Φυσικά έχετε φόβο γιατί θέλετε να είσαστε μια μονοπολική δύναμη. Θέλετε να έχετε την Ευρώπη η οποία θα είναι μαζί σας. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουμε τις καλές σχέσεις γειτονίας και την ειρήνη. Μια Ευρώπη η οποία δεν θα έχει την αμερικανική κυδαιμονία σας. Και με τρόπο επιθετικό. Γνωρίζετε πολύ καλά λοιπόν τη δική σας προπαγάνδα. Κύριε Πρέσβη, καλώς ήρθατε καταρχάς. Όντως είναι εξαιρετικές οι στιγμές που ζούμε σήμερα ψηφίζουν οι Ηνωμένες ε, με έναν ε, υποψήφιο ο οποίος δεν έχει καν καταθέσει τη φορολογική του δήλωση. Νομίζω ότι είναι πρωτοφανές αυτό και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες. Δεν θα πρέπει να ακολουθούν λαϊκιστές όπως ο Τραμπ ή κάποιους λαϊκιστές εδώ πέρα οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τον Πούτιν. Πιστεύετε ότι η Χίλαρη θα καταφέρει να αποκριθεί τελικά στα στοιχεία που πήρε από το θεματολόγιο του Μπέρνι Σάντερς, δηλαδή ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τους φορολογικούς παραδείσους, ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την έλλειψη φορολογικών ρυθμίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, που τελικά είναι φαινόμενα που οδηγούν τους πολίτες να μην δείχνουν εμπιστοσύνη στα θεσμικά μας όργανα, στα χρηματοπιστωτικά όργανα και στις κυβερνήσεις. Θεωρείτε ότι αυτό θα αποτελέσει μέρος του θεματολογίου συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό, εξίσου σημαντικό μετά άλλα στοιχεία τα οποία θίξατε. Ευχαριστώ. Well, lots of questions, and I know the all eager to hear. Πολλές ερωτήσεις και υπάρχουν και υπουργοί εδώ πέρα που θέλουν να ακούσουν τις απαντήσεις. Πάρα πολλές ερωτήσεις ακούστηκαν για, το, για τα φαινόμενα λαϊκισμού. Το ζήτημα αυτό είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό, κρίσιμο θα μπορούσαμε να απορρίψουμε όντως τη βία της ρητορική που χρησιμοποιείται, την όλη ιστερία που δημιουργείται από ορισμένου. Ορισμένοι αναφέρθηκαν σε μια πολιτική η οποία υπερβαίνει πια την αλήθεια και δεν χρησιμοποιεί καν πραγματικά στοιχεία. Και πραγματικά σοκαρίστηκα όταν είδα στον Ηνωμένο Βασίλειο μετά την απόφαση του Τεγματικού Δικαστηρίου ότι ορισμένε εφημερίδε τη χώρα και όχι μόνο κίτρινο τύπο αλλά και κάποιε, πώ να το πούμε, πιο mainstream εφημερίδε λέγανε, είχαν τίτλους ο αναφέρονταν στους δικαστές και λέγανε ότι είναι εχθροί του λαού. Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε από τον Λένιν, από τους Ναζί και αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή στον Ομένο Βασίλειο που είναι το προπύργιο της κοινή λογικής και της δημοκρατίας. Κάτι έχει συμβεί σαφώς. Και ο λόγος για τον οποίο το λέω αυτό είναι επειδή πρέπει να καταλάβουμε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού τι συμβαίνει πια με την πολιτική. Ας αναλύσουμε καλά τα πράγματα, ας αναλύσουμε καλά την κατάσταση και ας καταλήξουμε στα σωστά συμπεράσματα. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει το αφήγημά μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πραγματικά ποια είναι τα βαθύτερα αίτια της λαϊκής αυτής οργής και νομίζω ότι αναφερθήκατε εσείς σε ένα, Ο Μπέρνι Σάνταρς ήθελε να δει μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη στις εμπορικές, για παράδειγμα, διαπραγματεύσεις δικαιοσύνη στο πώς αντιμετωπίζουμε τις πολυεθνικές όταν φοροδιαφεύγουν. Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει πρόοδος προς αυτό χάρη στον ΟΣΑ και απομένει βέβαια να γίνει μια πολύ σημαντική εργασία για να έχουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς εμπορικής άμυνας και να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα συστήματα εμπορικά, τα οποία δεν λειτουργούν σωστά αυτή τη στιγμή ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στι ΗΠΑ. Οι άνθρωποι θέλουν να γνωρίζουν ότι κινούνται σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό κόσμο με απόλυτη δικαιοσύνη. Θεωρούν ότι το σύστημα είναι διεφθαρμένο. Αυτό λένε πάρα πολλοί υποστηρικτέ του Ντόναλτ Τραμπ. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε λοιπόν ότι συμβαίνει κάτι το θεμελιώδε. Παρακολουθούμε την όλη συζήτηση, ξέρουμε τι έγινε στη Βαλονία, Νομίζω ότι πολλά συνδέονται περισσότερο με εσωτερικά ζητήματα πολιτική του Βελγίου και όχι τόσο πολύ με την ίδια τη φύση της συμφωνίας αυτής. Είχα διαβάσει όλες τις δηλώσεις που γίνανε σε σχέση με την συμφωνία αυτή τη ΣΕΤΑ και οι περισσότερες δηλώσεις που γίνανε εδώ σε τοπικό επίπεδο στο Βέλγιο δεν είχαν πραγματικά να κάνουν με την ίδια την ουσία της συμφωνίας, με το διατακτικό του ίδιο της συμφωνίας. Σαφώς υπήρχαν κάποιες ανησυχίε οι οποίες δεν θα έπρεπε καν υφίστανται από την αρχή. Όσον αφορά τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους για το TTIP. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το ζήτημα αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά αν θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε. Πιστεύω θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε τις επραγματεύσεις υπό την Προεδρία Κλίντον. Πρέπει να δούμε πώς θα διευθετήσουμε το ζήτημα ESDS. Ξέρουμε όμως τι έγινε με την ΣΥΤΑ και γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, δυνατότητα αυτή ε, διαιτητικών δικαστηρίων. Για τη Ρωσία τώρα. Δεν απολογούμε πραγματικά για αυτά τα οποία είπα. Έχω ζήσει στη Ρωσία και ζήτησα, ε, έζησα μάλιστα και Σοβιετική Ένωση πριν τον Κορμπατσόφ. Ξέρω ότι θα πει ολοκληρωτικό καθεστώς. Και φοβάμαι ότι σιγά σιγά επιστρέφουμε πίσω στις μέρες αυτές, όπου μη κυβερνητικέ οργανώσεις πραγματικά καταστρέφονται, διαλύονται, και πραγματικά τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δεινά από πολιτική και οικονομικής πλευράς για τη Ρωσία. Επιστρέφουν σε μία εποχή πριν την εποχή του Κορμπατσόφ. Επομένω. αν θα ε, ουσιαστικά το δημοκρατικό δικό μα σύστημα με την κατάσταση της Ρωσίας όπου καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, προφανώς αυτό το απορρίπτω. Το απορρίπτω εντελώ. Και Απορρίπτω επίσης αυτό το επιπόθηκε ότι η Ρωσία δεν επηρεάζει ε, ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ή ακόμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αντίθετα ως προς τη δήλωση αυτή και το γνωρίζουμε αυτό. Και αυτό θα αποτελέσει μια πολύ μεγάλη κοινή μας πρόκληση. Νομίζω ότι από κοινού θα μπορέσουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Εμεί εδώ οι σύμμαχοι, οι φίλοι που βλέπω στην αίθουσα αυτή, πολλά περισσότερα πράγματα μπορούμε να κάνουμε από κοινού για να καταδείξουμε πραγματικά τι συμβαίνει. Ορισμένα είναι δημόσια, γνωρίζουμε τι συμβαίνει με το εθνικό μέτωπο τη Γαλλία, αλλά πάλι δεν έχουν βγει ακόμα στην επιφάνεια. Νομίζω λοιπόν ότι από κοινού μπορούμε προ τα έξω να βγάλουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν ξέρω ποιος θα νικήσει τις εκλογές, αλλά καταλαβαίνετε ότι η εξωτερική πολιτική θα είναι εντελώ διαφορετική ανάμεσα στους δύο υποψηφίους. Ο Ντόναλτ Τραμπ έχει πει θα κάνει πάρα πολλά πράγματα, ενδεχομένω να μην καταφέρει να κάνει, χάρη στο Κογκρέσο ή χάρη στο Σύνταγμα των ΗΠΑ που δεν θα το επιτρέψει, αλλά όσον αφορά για παράδειγμα την νομοθεσία για τα βασανιστήρια, όσον αφορά τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Μεξικό, όσον αφορά τη στάση του απέναντι στην Κίνα, τα όσα έχει πει για τη μη διάδοση των όπλων. Το ότι θα μπορούσαν κάποιες χώρες στην Ασία να έχουν πυρηνικά όπλα. Καταλαβαίνετε ότι αν συμβούν αυτά τα πράγματα προφανώς θα επηρεάσουν και εμάς και την Ευρώπη. Για την παγκόσμια στρατηγική αναφερθήκατε σε στρατό, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχετε μία τάση ιδιαίτερα αυστηρή όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας και της άμυνας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δαπανείτε περισσότερο για ζητήματα ασφάλειας και άμυνας. Είμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Θεωρούμε ότι λαμβάνονται αυτή τη στιγμή κάποια κάποιες θετικές αποφάσεις και είναι βάσιμες οι ανησυχίες που έχουν ακουστεί αυτή τη στιγμή όσον αφορά το μόνιμο αυτό στρατηγείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θεωρούμε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, ούτε είναι απαραίτητα αναγκαίο. Μα λένε όλο και περισσότερο ότι στόχο τη νέα αυτή πολιτική είναι να καταφέρετε να εντοπίσετε στο πλαίσιο τη ε, συνθήκη τη Λισαβόνα τι δυνατότητε πιο ενισχυμένη συνεργασία πιο ενισχυμένη συνεργασία από ορισμένα κράτη-μέλη, να καταφέρουν ορισμένα κράτη-μέλη να, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του ΝΑΤΟ και πραγματικά να καταφέρουν ορισμένες χώρες να δαπανίσουν περισσότερα χρήματα για πραγματικές στρατιωτικές ικανότητες και όχι τόσο πολύ για ζητήματα όπως ε, η μισθή, για παράδειγμα. Τώρα το αν το Ηνωμένο Βασίλειο ή οι Ηνωμένε Πολιτείε εντοπίζονται στα βαθύτερα αίτια τη κρίση στη Μέση Ανατολή, εκτενέστατη συζήτηση θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά α μην επικεντρωνόμαστε στο παρελθόν. Θεωρώ ότι το μέλλον βρίθει προκλήσεων και θα πρέπει να ασχοληθούμε πραγματικά με τα όσα συμβαίνουν εκεί. Βλέπουμε ότι στη Μοσούλη οι προσπάθειες απελευθέρωσης της χώρας είναι πολύ σημαντικές. Η Κύπρος είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, μια πρόκληση και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε φέτος να λύσουμε το πρόβλημα. Για ποιο λόγο η Ουκρανία είναι τόσο σημαντική. Είναι εδώ πέρα στην αδελφή μου και τους κοιτάω. Για πάρα πολλούς λόγους. Ένα λόγο όμως θα έθετα, κυρίως εξαιτία των αξιών μας οι αξίες οι οποίες πρεσβεύουμε. Είδα μια πολύ συγκινητική ταινία και ελπίζω ότι θα ξαναπροβλεφθεί. Winter on Fire ονομάζεται η ταινία αυτή. Και εκεί πέρα βλέπουμε νεαρούς Ουκρανούς οι οποίοι ε, κρατάνε στα χέρια τους την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνουν μάχη και πολλές φορές χάνουν τη ζωή τους ακόμα και στους δρόμους του Κιέβου γιατί είπανε, τόλμησαν να πούν ότι θέλουν να σταματήσει η διαφθορά, θέλουν να είναι σε θέση να επιλέγουν το μέλλον τους, θέλουν να επιλέγουν ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Λέγανε οι άνθρωποι αυτοί ότι ανήκουμε στην Ευρώπη και λέγανε ότι η Ουκρανία ανήκει στην Ευρώπη. Συγκινήθηκα πραγματικά βλέποντας την ταινία αυτή, γιατί οι άνθρωποι αυτοί πλήρωσαν το ίστατο τίμημα. Αν λοιπόν τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει «Α, κουραστήκαμε, δεν μπορούμε πλέον να σε υποστηρίζουμε οικονομικά και διπλωματικά, αυτό θα είναι καταστροφικό. Γιατί τότε ποιο ο λόγο ύπαρξη Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν μπορεί να προασπίσει τι αξίε τη και αν δεν μπορεί να προασπίσει χώρε που έχουν μια ευρωπαϊκή ιστορία όπω Ουκρανία και που θέλουν να έρθουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να σημειώσουμε τώρα μεγαλύτερη πρόοδο όσον αφορά τα κοινά μα προγράμματα μείωση τη διαφθορά. Θεωρώ ότι πολύ μεγάλη πρόοδο έχει ήδη γίνει. Το TTIP προβλέπει ένα νέο μηχανισμό για την αντιμετώπιση και αυτών των φαινομένων. Θεωρώ ότι είναι ένα σχέδιο επενδυτικό και εμπορικό το οποίο είναι πιο φιλόδοξο από τα προηγούμενα εμπορικά σχέδια που είχαμε και έχουμε σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο στα ρυθμιστικά αυτά κεφάλαια πώς νομοθετούμε, πώς καταλήγουμε δηλαδή σε ρυθμίσεις, προκειμένου οι κανονισμοί και οι ρυθμίσεις να είναι πιο ευθυγραμμισμένες στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και σε συγκεκριμένου κλάδους έπειτα προσπαθούμε να δούμε αν μπορούμε να μειώσουμε τις αποκλήσεις στους κανονισμούς μας για να μειώσουμε και τις δεινές επιπτώσεις. Όλες οι μελέτες του TTIP έχουν δείξει ότι τα τρία τέταρτα των πιθανών προβλημάτων μπορούν να επιληθούν μέσω της κανονιστικής ευθυγράμμισης. Νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα ζητήματα, όχι ένα ακόμα. Όσον αφορά το CSDP, την κοινή εξωτερική πολιτική, πολιτική ασφάλεια και το ΝΑΤΟ, προσπαθούμε να περάσουμε ένα μήνυμα προ το Λονδίνο, αλλά είμαστε σαφεί. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να διαμεσολαβήσουν προκειμένου να χωρίσει τελικά το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε καμία περίπτωση θέλουμε να αναλάβουμε το ρόλο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για ζητήματα ΝΑΤΟ και για ζητήματα κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια και οικονομικά ζητήματα, το Ηνωμένο Βασίλειο και μετά το Brexit να παραμείνει στενό συνεργάτη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ζητάμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει περισσότερο χώρο και χρόνο στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προκειμένου να μπορέσουν να καταλήξουν και αυτοί σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για την πορεία που θα ακολουθήσουν. Αν η Κλίντον θα δείξει μεγαλύτερη τώρα πυγμή, δεν μπορώ να σα το πω. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέποντας ότι η Ρωσία προσπάθησε να πειράσει την εκλογική διαδικασία κάνοντας hacking στα συστήματα τα εκλογικά τα οποία έχουμε στις ΗΠΑ, καταλαβαίνετε τι αυτό σημαίνει. Ο ίδιος ο Λευκός Οίκος και ο αντιπρόεδρος Biden κάναν συγκεκριμένε δηλώσεις προς αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία έχει ξεπεράσει τα όρια και έχουμε και υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους της Ρωσίας που ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο αυτό. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό. Σίγουρα έχουμε πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να καλύψουμε τα επόμενα χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δραματίζει σαφώς ένα καθοριστικό ρόλο και εφόσον τα αποτελέσματα των εκλογών είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να είναι για μένα, ελπίζω να έχω τη δυνατότητα να σας ξαναδώ πολύ σύντομα. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος Μπροκ. Νομίζω ότι είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για την παρουσία σας εδώ σήμερα και πιστεύω ότι μπορούμε να ελπίζουμε για τη συνέχιση της σχέσης μας, για την προς το κοινό συμφέρον και οι δημοκρατικές δυνάμεις. Δεν θα πρέπει να έχουν καμιά αμφιβολία ότι στο τέλος της ημέρας θα κερδίσουν πάντα και όταν πρόκειται για την ε, ενέργεια κατά του Πούτιν, ίσως μπορεί να σας δώσει πληροφορίες ο κ. Σαφχάζων για τα λεφτά που παίρνουν από τον κ. Πούτιν για να χρηματοδοτούν την, πορτο, την ε, προπαγάνδα, ε, προπαγάνδα τους. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και πιστεύω ότι μετά από μια μεταβατική περίοδο ελπίζω θα μπορέσουμε και πάλι να συζητήσουμε <clears throat> την σχέση μας μετά από τη στιγμή που θα γνωρίζουμε τις προτεραιότητες της νέας Αμερικανικής Προεδρίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Έχουμε μαζί μας την Ιβάνα Κλίμπους Τσιντσάτσε, η οποία είναι αντιπρόεδρος της Ουκρανικής Κυβέρνησης, αρμόδια για θέματα ευρωπαϊκής και ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης. Μας ενδιαφέρει πολύ, κυρία Υπουργέ, να ακούσουμε από τα δικά σας χείλη τα, την αποψή σας για το σχέδιο εταιρική σχέσης μεταξύ της Ευρώπης και της Ουκρανίας. Υπήρξε μια συνάντηση πριν, πριν από 10 μέρες στο Παρίσι, όπου είχατε λάβει και εσείς ε, ε, λάβει μέρος, καθώς και οι ηγέτες του κόμματό και ήταν παρόν και ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και φυσικά και εγώ ίδιο και εγώ εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο με τον οποίο έγινε η ανταλλαγή απόψεων σε αυτό τον κλειστό κύκλο πώς θα μπορέσετε να υλοποιήσετε τους ε, μηχανισμούς ελέγχου <clears throat> με την παρουσία και του διαμεσολαβητή του ε, Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο του Πατ Κόξ για τα θέματα αυτά της Ουκρανίας. Επομένως βγήκαμε από αυτήν τη συνάντηση με κάποια ελπίδα ότι μπορούν τα πράγματα να προχωρήσουν καλύτερα σε ό,τι αφορά την βελτίωση της κατάστασης του κράτους δικαίου στην Ουκρανία. Αυτή ήταν μια πολύ καλή εμπειρία και γι' αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να γνωρίσουμε με ποιο τρόπο μετά από την πρόσφατη συνάντηση στο Βερολίνο βλέπετε την ε, πρόοδο των ενεργειών αυτών. Και επίσης για τη δυνατότητα η αποστολή του ΟΑΣΕ να προχωρήσει στα θέματα αυτά. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν κατά την άποψή σας πώς έχουν προχωρήσει τα πράγματα και εάν είναι εφικτό ο πρόεδρος Πούτιν της Ρωσίας να πείσει τους φίλους του στον Τόν Μπάς να επιτρέψουν την παρουσία της αποστολής αυτής του ΟΣΑ, ο ΑΣΕ Ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχετε λοιπόν. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Μπρόκ. Σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθυνθώ σε αυτήν ε, την αξιότιμη το αξιότιμο ακροατήριο και στα μέλη Εθνικών Κοινοβουλίων και θα ήθελα να σας ενημερώσω για την κατάστασή μας, για το που βρισκόμαστε σήμερα όταν περίπου τρία χρόνια έχουν περάσει από την αρχή της ε, επανάστασης της αξιοπρέπειας. Σας εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε όσους υποστήριξαν την Ουκρανία σε διάφορες διεθνείς και εθνικές κονίστρες για την οικονομική και τεχνική βοήθεια που λαμβάνουμε σε αυτήν την εποχή μετασχηματισμού. Εδώ και τρία χρόνια, στις 21 Νοεμβρίου του 2013, άρχισε η Επανάσταση της Αξιοπρέπειας και Είχαμε επίσης και την Συμφωνία Σύνδεσης τρία χρόνια αργότερα. Νομίζουμε αυτό το έγγραφο το οποίο υπεγράφηκε και επικυρώθηκε από 27 από τα κράτη-μέλη είναι ένας, ένα φύλλο πορείας, ένας χάρτης πορείας για την αλλαγή και ένα θεματολόγιο τόσο για την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέτει επίσης πάρα πολλές προκλήσεις για μας. Για μας στην Ουκρανία δεν είναι απλώς ένα έγγραφο αυτό, είναι ένα σύμβολο, ένα σύμβολο και η σημαία της μάχης μας για την ελευθερία. Εμείς οι Ουκρανοί δεν είμαστε τόσο διαφορετικοί από τα άλλα έθνη, θέλουμε ειρήνη, θέλουμε ασφάλεια, θέλουμε ε, κάποιο επίπεδο καλής διαβίωσης, επίπεδο ζωής βιωτικό. Και τώρα προσπαθούμε επίσης να κάνουμε τους εταίρους μας να συμμετέχουν. Αυτό που ζητούμε από την Ευρώπη, ε, ζητούμε μια ευκαιρία. Γι' αυτό ε, είμαστε, μας ανισχύει τόσο πολύ η κατάσταση που εξελίσσεται τώρα με την μη επικύρωση της συμφωνίας από τις κάτω χώρες. Ζητούμε μια ευκαιρία, όχι επειδή νομίζουμε ότι απλώς ε, τη δικαιούμαστε, διότι πιστεύουμε στις αξίες, ε, στις υποσχέσεις, στην αξιοπιστία και η Ουκρανία έχει επιλέξει την Ευρώπη και τιμωρήθηκε επειδή επέλεξε την Ευρώπη. Ας μην διατηνόμαστε ότι αυτή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ουκρανία είναι μόνο θέμα Ουκρανίας και Ρωσίας, είναι θέμα όλων μας. Μπορούμε να μείνουμε στο περιθώριο ή να μείνουμε ενωμένοι και να επιδείξουμε αλληλεγγύη. Έχουμε πλήρη συνείδηση των ιδιαιτεροτήτων αυτής της κατάστασης στις ε, κάτω χώρες ε, ότι θα υπάρξουν σύντομα εκλογές και είναι λυπηρό που η Συμφωνία ε, Σύνδεσης που υποστηρίχθηκε τόσο πολύ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από Εθνικά Κοινοβούλια τώρα έχει να αντιμετωπίσει αδικαιολόγητη αντίθεση αλλά ε, ελπίζουμε ότι μετά είδαμε τις προτάσεις Πρωθυπουργού Γιούτ από τον Κοινοβούλιο ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση και είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να εργαστούμε στενά με όλες τις πολιτικές ομάδες, με όλους τους εκπροσώπους για να βρούμε μια λύση που θα ικανοποιήσει τις ανησυχίες της αντικειμενικές των κατοχωρών και ότι οι κόκκινες γραμμές που είναι σημαντικές για την Ουκρανία δεν θα τις περάσει κανείς και ότι δεν θα έχουμε επαναδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας Σύνδεσης. Δεν περιμένουμε τροπολογίες και βασιζόμαστε ε, σε μια κατάσταση μη διακρίσεων απέναντι στην Ουκρανία. Κάνουμε έκκληση σε όλες τις πολιτικές ομάδες και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε σε αυτό το εγχείρημα, ούτως ώστε στις ε, κάτω χώρες ε, να δεχθούν αυτή τη λύση που είναι αποδεκτή από τις 27 χώρες που έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν την Ουκρανία για να υλοποιήσει την Συμφωνία Σύνδεσης. Στην εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής όπως θα γνωρίζετε εμείς προσπαθούμε ε, με μια πολύ δύσκολη κατάσταση στο ανατολικό μέρος. Έχουμε συνεχιζόμενο πόλεμο. Υβριδικός πόλεμος τον ονομάζουμε, αλλά είναι θερμός πόλεμος με την Ρωσική Ομοσπονδία στη δική μας επικράτεια. Επίσης έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε, το, το μέτωπο ε, των δύσκολων μεταρρυθμίσεων αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Βλέπουμε ήδη τα αποτελέσματα μερικών από αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Ε, οι δραστηριότητες που έχει αναλάβει η χώρα, ε, έχουμε για την ενέργεια, για τον φορολογικό τομέα, τον τραπεζικό τομέα, για την γεωγραφική διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και του εφοδιασμού του ενεργειακού. Μερικοί αριθμοί τώρα. Η Ουκρανία το Μάρτιο 2014 είχε 10.000 δολάρια στο ταμείο της, τώρα έχει αποδείξει ότι έφτασε στο επίπεδο όπου τα μακροοικονομικά έχουν σταθεροποιηθεί. Στο τέλος του έτους θα έχουμε μια μικρή ανάπτυξη, 1%. Το επόμενο έτος έχουμε μια πρόβλεψη 3% οικονομική μεγέθυνση, δηλαδή η οικονομία μας γίνεται πιο υγιής και βρισκόμαστε στη σωστή πορεία, στο σωστό δρόμο. Έχουμε περικόψει το έλλειμμα το δημοσιονομικό κατά 5%. Έχουμε ε, καθαρίσει το τραπεζικό τομέα ε, όπου υπήρχε τρομερή διαφθορά στην Ουκρανία ε, και έχουμε κλείσει 82 τράπεζες. 82 τράπεζες έχουν εξαλειφθεί από το τραπεζικό οποίο Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα γίνεται υγιέστερο, καθαρότερο και πιο ζωντανό. Έχουμε αυξήσει το τιμολόγιο του ενεργειακού σε 100% τώρα δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ε, τιμή ενέργειας ε, για ε, τις οικογένειες, για τις μικρές μεγάλες επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά και τις αρχές της κρατικές. Κλείσαμε λοιπόν την ψαλίδα διαφθοράς που υπήρχε στην Ουκρανία όλα αυτά τα χρόνια από την ανεξαρτησία το 1991. Για πρώτη φορά η Ναυτογκάς γίνεται επικερδής στην Ουκρανία που δεν ήταν η περίπτωση μετά την ανεξαρτησία για όλα τα χρόνια. Ήταν μια εταιρεία που είχε, λάμβανε μεγάλη επιδότηση από το κράτος κάθε χρόνο. Ξέρω ότι όλοι ακούσατε για, το γεγονός εμείς έχουμε ε, περάσει στο πρώτο στάδιο ε, των ε, δηλώσεων και είναι ένα μέσο για να αυξήσουμε την ε, λογοδοσία των πολιτικών, των δημοσίων υπαλλήλων και ελπίζουμε ότι αυτό θα εξασφαλίσει την αυξημένη εμπιστοσύνη του κοινού απέναντι στους θεσμούς αυτούς, στις πολιτικούς και στους υπαλλήλους του δημοσίου έχουμε Έχουμε την υπηρεσία πρόληψης ε, της διαφθοράς που μπορεί να επαληθεύσει όλες τις πληροφορίες και στην περίπτωση που εντοπίζει κάποια κατάσταση που δεν συνάδει με τον Ουκρανικό νόμο πρέπει να παραπέμψει τις υποθέσεις αυτές στην υπηρεσία κατά της διαφθοράς. Και θα ήθελα να αναφέρω ότι η επανάσταση της αξιοπρέπειας ήταν θέμα επιλογής της δικαιοσύνης απέναντι στην αδικία. Ε, είναι σημαντικό το ότι κατορθώσαμε να έχουμε τις τροπολογίες τις συνταγματικές που ψηφίστηκαν ε, για τον δικαστικό τομέα και τώρα ο δικαστικός τομέας έγινε αποτελεσματικός από ε, τις 30 Σεπτεμβρίου και έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα σύστημα διαφανές ε, διαγωνισμών για την επιλογή νέων δικαστών που μπαίνουν στο σύστημα ε, και ε, να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε ένα σύστημα που ήταν πολύ διαφθαρμένο. Το, το, η διαφθορά, η καταπολέμησή της δεν είναι μόνο, δεν γίνεται μόνο με την δημιουργία θεσμών και μονάδων, αλλά κλείνοντας και τα κενά ε, στους κανονισμούς της χώρας μας. Μία, ένα από τα επιτεύγματα για τα οποία είμαστε υπερήφανοι και που έχει επιπτώσεις πάνω στη διαφθορά είναι από την 1η Αυγούστου χρησιμοποιούμε Έχουμε ηλεκτρονικό ε, σύστημα διαγωνισμών, δημοσίων διαγωνισμών που μέχρι το τέλος του έτους ε, θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε 16% των δημοσίων δαπανών και εκεί μπορούμε και καλύπτουμε τα ε, κενά. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό, θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υπέβαλε τα μέτρα, τα αυτόνομα εμπορίου για την Ουκρανία και ζήτησε την υποστήριξη των Ευρωπαίων βουλευτών στην ψηφοφορία εδώ στο Κοινοβούλιο, διότι πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι ένα άλλο κίνητρο για μας στην Ουκρανία ούτω ώστε να προωθήσουμε τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο θέμα το οποίο πάνω στο οποίο θα ήθελα να προσελκύσω την προσοχή σας είναι η απελευθέρωση των θεωρήσεων, η συμφωνία. Η Ουκρανία έχει 144 απαιτήσει που τέθηκαν για το σχέδιο δράσης απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Πρόκειται για μέτρα πάρα πολύ οδυνηρά τα οποία πρέπει ε, να λάβουμε. Και τώρα εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει. Χαιρόμαστε με την απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επίτροπη, την νομική διάταξη και χαιρόμαστε για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, της Επιτροπής ΑΦΕΤ και για τα μηνύματα τα οποία τέθηκαν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτάπετος και θα ήθελα να υπάρξει αυτή η δυνατότητα για ε, να μην είναι η Ουκρανία όμοιρος ενός τριμερούς ε, διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών ε, θεσμών για τον μηχανισμό αυτών. Ελπίζουμε ότι θα απελευθερωθεί το θέμα των θεωρήσεων. Είναι θέμα νομίζω αξιοπιστίας αν το ένα μέρος αποδίδει και παράγει αποτελέσματα νομίζουμε ότι και το άλλο μέρος θα πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία. Και εδώ με όλα τα σημάδια, τα θετικά που έχουμε από τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να αναλάβετε μέτρα και να υποστηρίξετε τους Ουκρανούς οι οποίοι ε, δικαιούνται πλήρως ε, να έχουν αυτό το προνόμιο, διότι κάνουν πολλά ως πολίτες, διότι τηρήσαμε τις ε, δεσμεύσεις μας. Ζούμε σε μια εποχή όπου μια άλλη πρόκληση η οποία ε, κάνει τις πόρους μας να παρεκκλίνουν από τον αρχικό του σκοπό. Έχουμε ανθρώπινους ε, πόρους επίσης που ε, διοχετεύονται προς τον, την διένεξη. Έχουμε μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού του ΑΕΠ που αφιερώνεται στην άμυνα. Έχουμε δει επίσης ότι το τίμημα θανάτων αυξάνεται των στρατιωτικών μας. Ε, βλέπουμε ότι όσοι έχουν εκπαιδευτεί από την Ρωσική Ομοσπονδία, πώς φέρονται βλέπουμε ότι έχουμε περιορισμούς ε, ε, των δραστηριοτήτων της ειδική αποστολής του ΟΑΣΕ ε, και έχουμε επίσης βλάβες στα τεχνικά μέσα. Αναφέρω 700 ε, άρματα ε, στο έδαφος του Ντομπάσα. Έχουμε επίσης συστήματα ρουκετών, βλημάτων, διάφορα εξαρτήματα που είναι επιπλέον των ρωσικών δυνάμεων που είναι παρούσες και που τις διαχειρίζεται η Ρωσική Ομοσπονδία σχετικά με τις διαπραγματεύσεις του Μίνσκ ε, και τις συνεδριάσεις ε, στο Βερολίνο, του σχήματος Νόρμαντι, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε για έναν χάρτη πορείας που θα έχει μια αλληλουχία για τις, τα διάφορα μέτρα, τις προϋποθέσεις, τα προαπαιτούμενα, τα ανθρωπιστικά που θα πρέπει να ικανοποιηθούν και μετά από αυτό θα μπορούμε να επανέλθουμε στην πολιτικό θεματολόγιο που, για το οποίο πολλά έκανε η Ουκρανία και νομίζω πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσε να κάνει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι αν ακούσουμε τις φωνές ε, που ζητούν ε, να ξαναρχίσουν οι σχέσεις, να ενταθούν οι σχέσεις, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι περιμένουμε από την Ευρώπη και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι είπε ο Τσέρτσιλ σε κάποιο σημείο μην, διαλέξετε την ντροπή, τον πόλεμο. Νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι δυστυχώς Είμαστε, ζητούμε ενότητα, αλληλεγγύη και όχι διχασμό. Ζητούμε ελεύθερη και ε, δημοκρατία. Πιστεύουμε στην ε, ελευθερία, στη δημοκρατία και θα πρέπει ε, να υποστηρίξουμε αυτές τις αξίες. Δεν πρέπει να προσπαθούμε να παίξουμε σκάκι με το Κρεμλίνο διότι θα πρέπει να φύγουμε όταν το επιθυμήσουν. Η Ουκρανία δεν διάλεξε την Ρωσία ως εχθρό. Η Ρωσία διάλεξε την Ουκρανία ως εχθρό. Δεν να είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποφάσισε η Ρωσία να είναι ο αντίπαλος της. Η Ρωσία διάλεξε την Ευρώπη ως αντίπαλο. Και εμείς θα τηρήσουμε τις αποφάσεις μας και θα εργαστούμε στη χώρα μας για να μπορέσουμε να γίνουμε μια καλύτερη χώρα, μια χώρα που θα έχει κανόνες, ε, κράτους δικαίου, διαδικασίες, ίδιες με τις χώρες που κατά τη γνώμη μας είναι επιτυχημένες και είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κλίμπους, θα συνεχίσω στα ισπανικά. Αρχίζει η συζήτηση με πρώτον ομιλητή τον κύριο Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ και καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήδη βρεθήκαμε στο Κίεβο την προηγούμενη εβδομάδα σε μια αποστολή της Προεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας και χαίρομαι για την ευκαιρία που είχατε να μας παρουσιάσετε την πορεία της Ουκρανίας και της προέδρου, της που επιτύχατε στην Ουκρανία. Είναι ήδη αξιοθαύμαστο για το πόσο, με πόση επιμονή μπορέσατε ως ε, δυνάμεις μεταρρυθμιστικές μπορέσατε να βγείτε από την προηγούμενη κατάσταση της Ουκρανίας και να οικοδομήσετε ένα πραγματικά φυσιολογικό και ομαλό κρατικό μηχανισμό. Αυτό αξίζει την επικρότηση και τον θαυμασμό σας. Μας. Ήμουνα στο Κίεβο την προηγούμενη φορά, <clears throat> την προηγούμενη εβδομάδα και είδαμε ότι εξακολουθούν Ρώσοι στρατιώτες να σκοτώνουν πολίτες της Ουκρανίας. Δεν πρέπει λοιπόν για πραγματιστικούς λόγους να αποκρύψουμε την αλήθεια, θα πρέπει να την αποκαλύψουμε αν πρόκειται να καταλήξουμε σε πραγματικές ε, αποφάσεις. Θέλω να εστιάσω στην ε, ελευθερία προξενικών θεωρήσεων, γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο για την Ευρώπη. Αφήνω το Κόσοβο και την Τουρκία κατά μέρο. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Γεωργία και η Ουκρανία είναι σημαντικέ χώρε, δεν τι αντιμετωπίζουμε σαν πακέτο. Αλλά <clears throat> με ενδιαφέρει αυτό που είπατε κυρία Υπουργέ. Είπατε ότι η Ουκρανία έχει εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις. Είναι σωστό αυτό. Και είναι απαραίτητο από τη δική μας πλευρά και εμείς να κάνουμε τα απαραίτητα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνει με αποτελεσματικό χαρακτήρα αυτό. Ο τριγωνικός διάλογος λοιπόν θα πρέπει να έχει σαν μοναδικό ε, ρόλο να υποστηρίξει την φιλελευθερωποίηση των προξενικών θεωρήσεων και όχι να την τορπιλήσει. Ο εισηγητής μας είπε ότι υπάρχει ένα σημείο μονάχα που δεν έχει υπάρξει συμφωνία και το οποίο έχει ε, αναβληθεί. Στις 24 Νοεμβρίου, που είναι η τρίτη ε, επέτειος του Ευρωμαϊντάν, έχουμε μία ε, διάσκεψη κορυφής Ευρώπης-Ουκρανίας δεν πρέπει όμως να χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση αμοιβαίων κατηγοριών γιατί υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να παρουσιάσουν την ε, προπαγάνδα ότι οι Ευρωπαίοι δεν αξιόπιστοι, δεν πρόκειται να αποδώσουν την ελευθερία θεωρήσεων και οι Ρώσοι είναι πολύ πιο αξιόπιστοι. Και εδώ είναι μια έκκληση και προς τους συναδέλφους από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που ασχολούνται με το θέμα αυτό να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό των προξενικών θεωρήσεων ώστε να μην είμαστε αναξιόπιστοι και στις 24 Νοεμβρίου. Αυτό είναι λοιπόν ένα, μια έκκληση που κάνω. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εξωτερικής πολιτικής που θα πρέπει εμείς να κάνουμε τα απαραίτητα για να βοηθήσουμε τις δυνάμεις μεταρρύθμισης στην Ουκρανία και όχι αυτούς οι οποίοι θέλουν να εμποδίσουν την πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος, Μάκερ, <clears throat> έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Κλίμπουτς. κύριο κύριος χαιρόμαστε που σας έχουμε και πάλι εδώ. Είμαι φίλος Ουκρανίας όπως ξέρετε έχω υποστηρίξει την Ουκρανία, έχω υποστηρίξει και την φιλελευθερωποίηση προξενικών θεωρήσεων, την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, την υπεράσπιση του εδάφους της έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έχουν γίνει λοιπόν πολλές μεταρρυθμίσεις και υπάρχουν και άλλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες επίκυνται. Για να είμαστε φίλοι πρέπει να πούμε και την αλήθεια όταν συζητάμε μεταξύ μας. Όταν βλέπω τις ειδήσει για την Ουκρανία δεν βλέπω πάντα ενθαρρυντικά μόνο νέα. Υπήρξαν απεργίες ανθρακορίχων γιατί φαίνεται ότι δεν έχουν πληρωθεί για πολλούς μήνες και επίσης έχουμε την ε, δήλωση στοιχείων ενεργητικού για τους πολιτικούς στην ε, Ουκρανία. Είναι ένα σύστημα που επιτέλους λειτουργεί, αλλά ο πληθυσμός νιώθει αγανάκτηση μετά από αυτά που βλέπει όταν βλέπει το πόσα αγαθά πολυτελείας που έχουν στα χέρια τους πολιτικοί, αυτό είναι κάτι το οποίο εντυπωσιάζει και αποτροπιάζει τους πολίτες της ε, Ουκρανίας. Είχαν ένα σύνολο σε στοιχεία ενεργητικού πάνω από ένα δισεκατομμύριο, όσο ήταν και το δάνειο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην <clears throat> ε, Ουκρανία. Όταν εγώ λοιπόν θέλω να υπερασπιστώ την Ουκρανία στου ενώπιον των πολιτών μου, των εκλογέων μου, δεν το βρίσκω εύκολο. Καλό είναι που υπήρξε αυτή η δήλωση αγαθών των πολιτών, αλλά αυτό δείχνει πόσο μεγάλη είναι η έκταση του προβλήματος της ε, διαφθοράς. Οι λίγοι εργαζόμενοι στο, στην υπηρεσία <clears throat> διαφθοράς θα πρέπει να αγωνιστούν για να καταλάβουν τι βρίσκεται πίσω από όλες αυτές τις ε, δηλώσεις. Ελπίζω λοιπόν ότι στο μέλλον θα μπορέσει να εμποδιστεί η άνθηση της <clears throat> διαφθοράς. Πρέπει οι πολίτες να αντιμετωπίσουν την διαφθορά που βρίσκεται σε επίπεδο καθημενο. Εγώ απλώς είχα στείλει ένα πακέτο στην Ουκρανία που είχε απλά πράγματα, κάποια αγαθά για το χειμώνα, ρούχα και ε, σοκολάτες και μου είπε ο συνομιλητής μου ότι θα έπρεπε να πληρώσει δασμούς 200 ε, ευρώ. Τελικά μόνο για να πάνε το πακέτο έπρεπε να πληρώσουν 75 ευρώ και μόνο. Εγώ πραγματικά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο με εξοργίζει. Δεν υπήρξε καμία ε, <clears throat> εξήγηση για όλα αυτά. Ουσιαστικά οι τελωνικές αρχές είναι κράτος εν κράτη. Και η μεταρρύθμιση στον τομέα αυτών των τελωνιακών θεμάτων ήταν, μια από τα προ... ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα για την φιλελευθερωποίηση προξενικών θεωρήσεων. Αλλά οι απλοί άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται αυτή τη διαφθορά σε καθημερινό επίπεδο. Τι κάνετε για όλα αυτά. Όσο δεν γίνεται κάτι τέτοιο, δεν θα έχετε την εμπιστοσύνη του λαού στην Ουκρανία. Εγώ υποστηρίζω λοιπόν τη φιλελευθερωποίηση της, ε, το προψηφιακό θεωρήσεων και θα το συνεχίσει να το κάνει η κυβέρνησή μου. Αλλά εξακολουθώ να αγωνίζομαι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ουκρανία, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορείτε να κάνετε και εσείς να μας βοηθήσετε σε αυτόν τον αγώνα. το Σαστοεβίτσιος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Κυρία Κλίμπουτς, καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντα είναι ιδιαίτερη χαρά να σας βλέπουμε, γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι έχετε αφοσιωθεί στη συνεργασία αυτή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας. Ως μέλος της, του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας, είχατε ασχοληθεί ιδιαίτερα και με τα ζητήματα σύνδεση μεταξύ Ουκρανία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ λοιπόν ότι είστε ο πλέον κατάλληλο άνθρωπο για να απαντήσει στι ερωτήσει που ενδεχομένω εμεί να έχουμε. Οι δικέ μου ερωτήσει είναι οι ακόλουθε. Πρώτον, ποια είναι η επιρροή από τη ροή πληροφοριών ή την προπαγάνδα που προέρχεται από τη Ρωσία και κατευθύνεται προς την Ουκρανία. Η πλειονότητα των πολιτών της Ουκρανίας προφανώς καταλαβαίνουν ρωσικά. Το να προβάλλονται λοιπόν τα μηνύματα αυτά νομίζω ότι επηρεάζεται τόσο η άποψη των Ουκρανών όσο πολλές φορές και η συναισθηματική τους τελικά κατάσταση. Ε, τι θα είχατε να πείτε για παράδειγμα για, τους, για τα κανάλια εκείνα τα οποία χρηματοδοτούνται από τη Ρωσία και λειτουργούν στην Ουκρανία. Βλέπουμε ότι ε, η ρωσική πλευρά καταβάλει όλο και περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να έρθει σε επαφή με την ουκρανική πλευρά. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συντάξουμε μια ειδική έκθεση για ζητήματα προπαγάνδας και παραπληροφόρησης που συμβαίνει βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που προέρχεται από διάφορες πλευρές και όχι μόνο από τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ομοφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί δεν θεωρούν ορισμένοι ότι η προπαγάνδα αυτή που προέρχεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει τελικά τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αφήγημα πάντως που προωθεί η Ρωσία ενδεχομένως να επηρεάζει ακόμα και τα ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ουκρανία και κάτι αντίστοιχο θα ίσχυε ουσιαστικά για οποιαδήποτε ελεύθερη δημοκρατία. <coughs> Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το ζήτημα αυτό που έχει να κάνει με τις ηλεκτρονικές δηλώσεις. Εγκρίθηκε το σύστημα αυτό, σας συγχαίρω πραγματικά και όντως αποκάλυψε πάρα πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα αυτή η ηλεκτρονική δήλωση των περιουσιακών στοιχείων. Από ό,τι φάνηκε πάρα πολύ αξιωματούχοι, είναι πολύ πλούσιοι και θα μπορούσαν οι ίδιοι μέσω της προσωπικής τους περιουσίας να υποστηρίξουν τελικά την ουκρανική οικονομία αγοράζοντας για παράδειγμα ομόλογα ουκρανικά τα οποία θα εξέδιδε η κεντρική σας τράπεζα και κατά αυτόν τον τρόπο θα χρηματοδοτούσαν έργα υποδομής και άλλα έργα στην Ουκρανία. Το ερώτημά μου είναι το ακόλουθο. Ποια ήταν η αντίδραση ακριβώς του πληθυσμού στη χώρα σας όταν βγήκαν στην επιφάνεια όλες αυτές οι πληροφορίες, όταν κοινοποιήθηκαν, ποια ήταν η αντίδραση του κοινού εν γέννη όταν χρειάστηκε ότι ό, να παραδεχθούν όλοι αυτοί οι πολιτικοί ότι είχαν μια τεράστια τελικά περιουσία στα σπίτια τους τελικά κρυμμένη, όχι απαραίτητα μέσω τραπεζικών καταθέσεων και ούτε μέσω συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Πρόκειται κυρίως για μετρητά, μύθιτη περιουσία που είχαν και κρατούσαν στο σπίτι τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπρόεδρε της ε, Ουκρανίας για τα σαφή σας λόγια. Αν τώρα <clears throat> βλέπετε να υπάρχουν επικρίσεις κατά της ε, Ουκρανίας, θέλω να σου υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι το σοβιετικό σύστημα βασιζόταν στην διαφθορά και χρειάζονται πολλά χρόνια για να ξεπεραστεί αυτό το σύστημα. Εγώ θέλω να εκφράσω την, το θαυμασμό μου για αυτά τα οποία έχετε κάνει στη χώρα σας σε ό,τι αφορά τη φιλελευθερωποίηση για τις προξενικές θεωρίες, θέλω να σταθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Γκάλερ, τον οποίο υποστηρίζω ε, απόλυτα. Και έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα για σας. Πρέπει να πω <clears throat> ότι ήδη πριν από την επίσκεψή μου στην Ουκρανία την προηγούμενη εβδομάδα είχα επηρεαστεί από την ρωσική προπαγάνδα. Αλλά είδα ότι πάρα πολλά πράγματα είναι διαφορετικά από την ρωσική προπαγάνδα, χάρη και στη δική μου συνάντηση μαζί σας. Μήπως θα ήταν δυνατό η Ουκρανική πλευρά να δίδει και περισσότερες πληροφορίες προς τον τύπο ώστε να μπορέσει να αποτελέσει ένα αντίβαρο στην ρωσική προπαγάνδα. Αυτό είναι πάρα πολύ αποφασιστικό και <clears throat> αν άτομα σαν και εμένα είχαν επηρεαστεί από αυτή την προπαγάνδα, πρέπει και εσείς να κάνετε πολύ περισσότερο για να την αντισταθμίσετε. Ο κύριο Σουάσεμερ από το Τσεχικό Κοινοβούλιο έχει το λόγο. Mm. μάλλον, η ορισμένα σχόλια για την Ουκρανία έχει επικριθεί η διαφθορά στην Ουκρανία, ελέγχθη σωστά ότι η Ουκρανία ήταν τμήμα του Σοβιετικού συστήματος. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε όμως ότι κάποιοι πρώην πρόεδροι της Ουκρανίας με την υποστήριξη της Ρωσίας χρησιμοποίησαν τη διαφθορά για να υποστηρίξουν το δικό τους σύστημα. Εμείς πρέπει να υποστηρίξουμε την Ουκρανία όχι μονάχα γιατί έτσι θα υπερασπιστούμε την Ευρώπη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την κατάληψη ενός εδάφους μιας ευρωπαϊκής χώρας να γίνει τμήμα του ρωσικού συστήματος. Πρέπει να κατανοήσουμε όμως το εξής. Αν η Μόσχα καταφέρει να πάρει την εξουσία πάνω από το Κίεβο, τότε θα γίνει σαφές ότι μετά από την σταδιακή απόσυρση των Αμερικανικών στα, στρατευμάτων από την ε, Ευρώπη και τη μεταφορά τους στον Ειρηνικό θα είναι σαφές ποιος θα είναι ο κυρίαρχος της Ευρώπης στον 21ο αιώνα. Αυτά θέλει ο Πούτιν. Δεν θέλει μόνο αμερικά χωριά στην Ανατολική Ουκρανία και τη βιομηχανία του Ντόνιετσκ. Δεν θέλει αυτό. Θέλει όλη την Ουκρανία γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έχει τη δυνατότητα να είναι ο κυρίαρχος και ο επικυρίαρχος όλης της Ευρώπης. Αυτό θέλει. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι η Ουκρανία είναι μια χώρα που έχει το μέγεθος της Γαλλίας και ένα σχεδόν συγκρίσιμο πληθυσμό. Είναι μια πλούσια χώρα. Μια πληροφορία που δεν πήραμε από σας κυρία μου είναι η εξή. Εγώ πήγα στην Ουκρανία πολλές φορές και ήταν πολύ ενθαρρυντικά το να δούμε την κοινωνία των πολιτών που λειτουργεί εκεί και έτσι έχουμε μια πρόσφατη εξέλιξη που έχει λάβει η χώρα. Βλέπουμε ότι η κοινωνία των πολιτών έχει εκφράσει την απόψή της και είναι πολύ δυναμική. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς για το γεγονός ότι κατάφερε με τον τρόπο αυτό να ξαναφέρει κοντά τους Ουκρανούς στην κυβέρνησή τους βλέπουν ότι η Ουκρανία είναι η πατρίδα τους και επίσης καταφέρει να αφυπνίσει την κοινωνία των πολιτών. Παρόλα όλα αυτά τα προβλήματα και εγώ έχω πάει στα σύνορα μεταξύ Ουκρανίας και κατεχομένων εδαφών και είδα τα βομβαρδισμένα κτίρια, είδα τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν υποφέρει. Η Ουκρανία αγωνίζεται και για το καλό της Ευρώπης και η Ευρώπη πρέπει να την βοηθήσει γιατί μέχρι τώρα δεν έχει πραγματικά δείξει αλληλεγγύη. Έχουμε δύο ακόμα μιλητές, θα τους παρακαλέσω να είναι σύντομοι για να μπορέσει και η καλεσμένη μας να έχει 10 λεπτά. Ο κύριος Γιούρεκ. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είχαμε σήμερα, τη... τη χαρά κύριε Πρόεδρε να ακούσουμε σημαντικές δηλώσεις από την κυρία Μογκερίνη και από τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών και ιδιαίτερα για θέματα του, των εμπορικών σχέσεων με την Ουκρανία και την ασφάλεια εφοδιασμού ενέργεια. Πρόκειται και για τον αγωγό Nord Stream 2. Θέλω να σας ε, Υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αγωνιστεί εναντίον αυτή τη εξέλιξη. Δεν θέλουμε η στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας να ενισχυθεί με την οικονομική απομόνωση της Ουκρανίας. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε ούτε χθε ούτε σήμερα. Έχουμε και την, Έχουμε και την επέτειο, είχαμε πρόσφατα την επέτειο της ε, κατάληψης εξουσίας από τους Μπολσεβίκους πριν από 99 χρόνια. Ένα πραγματικό εφιάλτη. Το τελευταίο ε, μνημείο στο Λένιν μόνο πρόσφατα εξαφανίστηκε στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι σημαντικό μόναχα για τη δική σας ιστορία, αλλά είναι και ένα πολύ καλό μήνυμα για την Δύση και την Ευρώπη. είσαστε μια πρωτοπορία στην Ουκρανία και σε ό,τι αφορά την ιστορία δεν έχουμε να σας δώσουμε κανένα δίδαγμα και μήνυμα. Αλλά θα πρέπει να τονίσω ότι θα πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα για την αποσοβιετικοποίηση της ε, ε Ουκρανίας. Πρέπει να επαναφέρουμε και το, το ναό του το όπου είχε καταστραφεί και είχε πάψει να λειτουργεί σαν εκκλησία. Υπάρχει η εκκλησία της Μαρίας Μαγδαλένας που είχε χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς και από ότι για εκκλησία. Θα πρέπει να ξαναλάβει το χαρακτήρα της και αυτό θα είναι σημαντικό για την Ουκρανία. Η κυρία Καλνιέτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια παρουσίαση ολοκληρωμένη σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, την διαδικασία μεταρρυθμίσεων, τα επιτεύγματα και τα προβλήματα που έχετε. Κάθε φορά διαβάζω άρθρα στο Economist, τόσο καλό περιοδικό, για τις μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι είναι μόνο, μόνο δύο χρόνια από τότε που η Ουκρανία ασχολείται με, τον, με τις μεταρρυθμίσεις, ακολουθεί το δρόμο των μεταρρυθμίσεων σε περιοχή όπου υπάρχει πόλεμο στην επικράτεια της Ουκρανίας. Και νομίζω ότι η ρωσική προπαγάνδα το, τη πλήση εγκεφάλων των Ευρωπαίων διανομένων, είναι πάρα πολύ δυνατές. Δεν έχουν καμία έννοια ε, της πραγματικότητας, της αλήθειας. Είμαι σε χώρα που πέρασε από το δρόμο των μεταρρυθμίσεων και ακόμα δεν τις έχουμε ολοκληρώσει. Σήμερα στην Ουκρανία είναι το πρόβλημα της κοινωνίας των πολιτών που δεν δέχεται να επανέλθει εκεί που βρισκόταν ε, πριν από το Μεϊντάν. Και λυπούμε που η απελευθέρωση των θεωρήσεων έχει ε, μείνει στάσιμη και έχει ανασταλεί και το θέμα της σύνδεσης. Είναι θέμα αξιοπιστίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να βρούμε αποτελέσματα. Το διάλογος πρέπει να βρει τον τρόπο να υπερνικήσουμε τα εμπόδια για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Θα έχω δύο ερωτήσεις να σας θέσω, κυρία Αντιπρόεδρε. Πρώτον, ε, σχετικά με το Nord Stream 2. Πώς αξιολογείται τις ε, επιπτώσεις πάνω στον ενεργειακό τομέα στην Ουκρανία. Και η δεύτερη μου ερώτηση σχετίζεται με την βοήθεια που παρέχεται διαμέσου του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλειά σας, για τον τομέα της ασφαλείας σας. Ε, αποστολή συμβουλευτική για μεταρρυθμίσεις. Θεωρείτε ότι είναι αποτελεσματική αυτή η βοήθεια και ρεαλιστική ε, για τις ανάγκες σας. Είναι κατάλληλη για τις ανάγκες σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Μπόξκορτ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που μπορώ να σας χαιρετήσω εδώ, να σας ε, καλωσορίσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ουκρανία. Σας συγχαίρω για το περιεχόμενο της παρουσίασής σας. Ενημερωθήκαμε για τις προόδους ως προς την απελευθέρωση των θεωρήσεων θα ήθελα να τονίσω ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων βουλευτών υποστηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία και όχι μόνο με τρόπο συμβολικό, αλλά κατά τη γνώμη μας η Ουκρανία θα έπρεπε το συντομότερο δυνατόν να επιτύχει αυτή την απελευθέρωση, διότι πληρεί όλες τις απαιτήσει, όλα τα προαπαιτούμενα, τα κριτήρια και τώρα δεν μπορούμε να αναβάλουμε αυτή την απόφαση η κυβέρνηση ε, τόνισε επανελειμμένα αυτήν την αναγκαιότητα. Χαιρόμεθα που η Ουκρανία είναι υπέρ της Ευρώπης, που στράφηκε στην Ευρώπη. Οι μειονότητες ε, στην Ουκρανία αντιπροσωπεύουν αυτήν την γνώμη. Και είναι κοινό μας συμφέρον να μπορέσετε να ακολουθήσετε την ευρωπαϊκή πορεία και να μπορέσουμε να μοιραστούμε αυτή την ίδια οδό. Θα ήθελα όμως να σας θέσω μία ερώτηση. Σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις ε, στο σύστημα της παιδείας, ε, της εκπαίδευσης, μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν τα δικαιώματα των μειονατήτων στο σύστημα το εκπαιδευτικό. Τι γίνεται με τις μεταρρυθμίσεις που προβλέπετε, μπορούν να τροποποιηθούν, πώς μπορούμε να τις επηρεάσουμε και να μεριμνήσουμε ούτως ώστε αυτή η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση να φτάσει σε καλό αποτέλεσμα. Ο κύριος Ρουσμπόλσκι, τελευταίος παρεμβαίνων. Ευχαριστώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την Ουκρανία που παραμένει ενωμένη στην ευρωπαϊκή της πορεία με θάρρος, διότι δεν υπάρχει άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρώπης που σε εποχή πολέμου προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις όπως εσείς. Δεχτείτε από μένα τρεις συγγνώμες, από μένα εκ μέρους πολλών εδώ. Πρώτα απ' όλα διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατάει όμοιρο την Συμφωνία ε, Σύνδεσης λόγω του ξενοφοβικού διπομψηφίσματος στις κάτω χώρες. Μας συγχωρείτε. Δεύτερον, για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην απελευθέρωση των θεωρήσεων ε, που είναι όμοιρος, αν θέλετε, της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Συγγνώμη. Και μια τρίτη συγγνώμη. Λυπούμε διότι δεν επιλύουμε όπως θα έπρεπε το πρόβλημα του Nord Stream 2 και, και για το OPAL που είναι το μισό απομονώνοντας από ενεργειακής πλευράς και από πλευράς ασφαλείας ε, την ε, Ουκρανία ε, που έχει πολιτικό, πολιτικά συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Μας συγχωρείτε. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην προσκεκλημένη μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω με την τελευταία παρατήρηση του κυρίου Σάριους Βόλφσκι. Σας ευχαριστώ που θίξετε το ζήτημα του ΟΠΑΛ, γιατί όντως συνδέεται μετά όσα είπαμε για το North Stream και θεωρούμε ότι τελικά είναι ένα πολιτικό κυριοσχέδιο το οποίο δεν είναι οικονομικά βιώσιμο ούτε οικονομικά δικαιολογούμενο τελικά προτάθηκε μεταξύ άλλων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ε, δεν θα απαιτείται πλέον η διαμεσολάβηση της Ουκρανίας ή τουλάχιστον ότι η Ουκρανική επικράτεια δεν θα είναι πλέον χώρος διαμετακόμισης και διέλευσης για το φυσικό αέριο. Μία ακόμη απόπειρα δηλαδή παράκαμψης της Ουκρανίας. Όσον αφορά τώρα την απόφαση που λήφθη για τον ΟΠΑΛ, θα έλεγα ότι ήταν αναπάντεχη η απόφαση αυτή, γιατί εμεί θεωρούσαμε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα και όλη η σχετική ενεργειακή δέσμη είχε να κάνει τελικά με την αλληλεγγύη και ότι δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να επιτρέπει δραστηριότητες οι οποίες θα έβαλαν κατά του ανταγωνισμού και ακριβώς αυτό τελικά έγινε με την απόφαση για τον αγωγό ΠΑΛ. Ελπίζω ότι θα καταφέρετε με κάποιο τρόπο να ανατρέψετε την απόφαση αυτή και να βρεθεί τελικά μια εναλλακτική λύση. Κατά αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι απάντησα τόσο για το North Stream 2 και για τον ΟΠΑΛ. Και σχετίζεται επίσης αυτό με αυτό που είπε η κυρία Κανιέτε πριν από λίγο, το ότι η Gazprom έχει τελικά μία δεσπόζουσα θέση, την οποία προσπαθεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο ουσιαστικά προσπαθεί να καταχραστεί ακόμα περισσότερο και μέσω του ΟΠΑΛ την θέση της. Ουσιαστικά δεν έχει να κάνει καθόλου με κάποια οικονομική στρατηγική, ούτε εξυπηρετεί πραγματικά οικονομικά συμφέροντα, ούτε συνάδει βέβαια με ένα θεμητό οικονομικό ανταγωνισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιούρεκ που ε, αναφερθήκατε στο ότι ε, προσπαθούμε να επιστρέψουμε κάπως στις ρίζες μας. Όπως είπε πριν από λίγο και ο Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος είπε ότι έζησε στη Σοβιετική Ένωση και εγώ μπορώ να πω ότι έχω ζήσει στη ε, Σοβιετική Ένωση και θυμάμαι πάρα πολύ καλά πώς η συναγωγή, η εκκλησία της περιοχής μου γίνανε αποθήκες ή γίνανε θέατρα για μαριονέτες κτλ. Σαφώς η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σήμερα. Σαφώς δεν θέλουμε μία σοβιετικοποίηση της χώρας μας. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι σεβόμαστε πολύ περισσότερο τις διαφορετικές θρησκείες και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είμαστε ένα έθνος, μια χώρα πολλών διαφορετικών εθνοτήτων. Και όσον αφορά τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην Ουκρανία, τα τηρούμε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μία τρανή απόδειξη είναι για παράδειγμα η ουγγρική μειονότητα στην Ουκρανία, η οποία συμμετέχει σε ένα περιφερειακό συμβούλιο. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι και στο πολιτικό προσκήνιο είναι δυνατόν να εκπροσωπηθούν όλες οι μειονότητες και ότι δεν προβλέπονται αποκλεισμοί. Όσον αφορά τώρα την προπαγάνδα που προέρχεται από τη Ρωσία, ετέθη ένα σχετικό ερώτημα. Ξέρετε ότι η ρωσική προπαγάνδα είναι η εξή ότι ήρθαν για να προστατεύσουν τους α, Εγώ ε, προέρχομαι από το Κίεβο, μεγάλωσα στο Κίεβο και όταν ένα σχολείο, ένα 80% των συμμαθητών μου μιλούσαν στο σπίτι τους ρωσικά. Όχι επειδή ήταν ε, ρωσόφωνοι λόγω των γονιών τους ή των παππούδων και των γιαγιάδων τους, ήταν του σειρμού εκείνη την εποχή να μιλά κανείς ρωσικά. Προσπαθούσαν να δείξουν ότι προσαρμόζονται πιο αποτελεσματικά στο καθεστώς Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν μια προσπάθεια, αν θέλετε, προσαρμογής από τους ανθρώπους εκείνους που ήθελαν να επιτύχουν μετά από 20-25 χρόνια τα δικά μου τα παιδιά πλέον πηγαίνουν στο σχολείο, στο κέντρο του Κιέβου, εκεί που σπούδασα και εγώ και πάλι στην τάξη τους είναι από τα ελάχιστα παιδιά τα οποία μιλάνε ουκρανικά για παράδειγμα κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων. Επομένως, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει καμία απολύτως απειλή όσον αφορά την χρήση της ρωσικής γλώσσας στο Κιεβό ή οπουδήποτε αλλού στην Ουκρανία. Δεν υφίσταται τέτοιο κίνδυνος, δεν υφίσταται τέτοια απειλή. Είναι ένας μύθος που χρησιμοποίησε η Ρωσία στα πλαίσια της προπαγάνδας, προπαγάνδας της. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, τέτοιος κίνδυνος και τέτοια απειλή κατά της χρήσης της ρωσικής γλώσσας δεν υφίσταται στην Ουκρανία. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ε, ηλεκτρονικές και έντυπες εφημερίδες, τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς, θέατρα, τα οποία χρησιμοποιούν πολλές διαφορετικές γλώσσες και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει καμία απολύτως απειλή κατά της χρήσης ε, της ρωσικής γλώσσας. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένας από τους μύθους, ένα από τα ψέματα που χρησιμοποιεί η ρωσική προπαγάνδα η οποία ναι όντως ανταποκρίνεται και προσπαθεί να κεντρήσει το ενδιαφέρον των Ουκρανών. Πριν από λίγο, δεν κάνω λάθος, ένας Ευρωβουλευτής πήρε το λόγο και είπε ότι από οικονομική πλευρά οι άνθρωποι εξακολουθούν και υποφέρουν. Όντως η μακροοικονομική σταθεροποίηση δεν μεταφράζεται μία ανοιχτή σε ευημερία για τον καθένα από τους πολίτες της Ουκρανίας. Παράλληλα όμως είναι πάρα πολύ εύκολο για μια χώρα η οποία συναισθηματικά και οικονομικά βρίσκεται σε ύφεση, είναι καταπονημένη αν θέλετε, είναι πολύ εύκολο για κάποιον να αναμοχλεύει όλα αυτά τα εθνικιστικά πάθη, να αναμοχλεύει όλη αυτή την εθνικιστική ρητορική η οποία υπόσχεται παραδείσους και η οποία στην πραγματικότητα παραπλανά τους πολίτες. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι και πολλοί γείτονέ μας παίζουν το παιχνίδι αυτό για να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα. Και βέβαια θα μπορούσαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πούτιν, όχι μόνο γιατί ενίσχυσε το ηθικό των Ουκρανών πολιτών, αλλά γιατί δημιούργησε τελικά ένα πολιτικό έθνος γινόμαστε ένα πολιτικό έθνος ακριβώς επειδή πρέπει να κινητοποιηθούμε, ακριβώς επειδή πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να συμπληρωθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τονεί το σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην Ουκρανία. Με ιδιαίτερη περηφάνεια είμαι εκπρόσωπος της κοινωνίας των πολιτών στην κυβέρνηση της Ουκρανίας. Όλη μου τη ζωή έχω εργαστεί σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις και σε οργανώσεις εκπροσώπησης τη κοινωνίας των πολιτών. Και μπορώ να σας πω ότι μετά την επανάσταση της αξιοπρέπειας, μεταξύ άλλων, αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν να εργαστούν στην κυβέρνηση ήταν άνθρωποι σαν και εμένα που εργάζονταν σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Γιατί είπαμε ότι ακριβώς η μελλοντική μας κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε πολύ στενές σχέσεις και στο μέλλον με την κοινωνία των πολιτών. Τα θεσμικά όργανα της Ουκρανίας έπρεπε να μείνουν σε επαφή με τους πολίτες Ουκρανίας. Ακριβώς αυτό θέλαμε να διασφαλίσουμε. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα. Όσον αφορά τώρα τον πλούτο αυτό, το πόθεν έσχεστο το οποίο δηλώθηκε ηλεκτρονικά από τους αξιωματούχους της κυβέρνησης. Δεν θα μπορούσα βέβαια να πω ότι ενέκρινε τις αποκαλύψεις αυτές η κοινωνία της ε, Ουκρανίας. Προφανώς αυτό δεν χαροποίησε τους πολίτες. Πολλοί περίμεναν να δούνε τελικά τι θα αποκάλυπταν οι ηλεκτρονικές αυτές δηλώσεις, είδανε τις αποκαλύψεις αυτές, αλλά βρισκόμαστε μόνο στην αρχή της όλης διαδικασίας, δεν το τέλος διαδικασίας. Καταρχάς σκεφτείτε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατον πριν από μερικά χρόνια. Το να δηλωθούν επισήμως, ηλεκτρονικά, στη ιστοσελίδα, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτικών αξιωματούχων θα ήταν αδιανόητο πριν από μερικά χρόνια. Αυτό λοιπόν αποτελεί ένα πρώτο μόνο βήμα ισχυρότερης λογοδοσίας. Και βέβαια ο απότερος στόχος είναι να αποδείξουν οι πολιτικοί αυτοί πώς απέκτησαν αυτή την περιουσία. Αν την απέκτησαν με αθέμητο τρόπο, αν μπορούν να δικαιολογήσουν την ύπαρξη αυτής της περιουσίας. Εκεί ακριβώς θα επικεντρωθεί το έργο της υπηρεσίας πρόληψης ε, της διαφθοράς. Είπατε ότι 300 άτομα, 300 πάλι θα χρειαστούν για να κάνουν τις επιθεωρήσεις αυτές. Μα μην ανησυχείτε, όλος ο λαός είναι από πίσω τους. Όλος ο λαός θα βοηθήσει προκειμένου να γίνει η ανάλυση αυτή. Στο παρελθόν όταν γίνανε οι δηλώσεις αυτές, είχαμε περίπου 3,5 εκατομμύρια επισκέψεις από τους πολίτες στην ιστοσελίδα. Και αυτό δεν ήταν επειδή οι πολίτες ήθελαν σώνει και καλά να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση, ήταν επειδή οι ίδιοι πολίτες ενδιαφέρονταν πολύ περισσότερο και θέλαν να δούνε πώς εξελίσσεται η διαδικασία. Είναι δικαίωμα των πολιτών να μπορούν πραγματικά να γνωρίζουν τα στοιχεία αυτά και η υπηρεσία πρόληψης διαφθοράς θα πρέπει προφανώς να λάβει δράση για όλες αυτές τις περιπτώσεις που ανέδειξε είτε η κοινωνία των πολιτών, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για συγκεκριμένα άτομα πολιτικού ή μέλη του Κοινοβουλίου. Έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα και προφανώς οι ελεγκτές αυτοί έχουν και την υποστήριξη του Ουκρανικού λαού όπως σας είπα. Επίσης, να ευχαριστήσω όλους όσοι μας υποστήριξαν και είπαν ότι θα πρέπει πραγματικά να προχωρήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο με την απελευθέρωση των προξενικών θεωρήσεων. Πραγματικά βασίζομαι σε εσά, τους ευρωβουλευτές. Εσείς ήσασταν οι πραγματικοί φίλοι και σύμμαχοί μας, οι πραγματικοί μας υποστηρικτές και ο διάλογος που έχω μαζί με εσά με την πρώην μου ιδιότητα ως ε, βουλευτής ήταν ένας διάλογος πάρα πολύ χρήσιμος, ήταν ένας ανοιχτός διάλογος, ένας διαφανής διάλογος και ένας διάλογος που ε, διέπεται από εμπιστοσύνη. Και θεωρώ ότι εξακολουθούμε και έχουμε αυτό το πνεύμα θετική συνεργασία και εμπιστοσύνη μεταξύ ημών και θεωρώ ότι μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο. Κύριε Ντεσμάκερ, αναφερθήκατε σε κάποιε περιπτώσει ε, συγκεκριμένες Είπατε, αναφερθήκατε σε ένα δέμα το οποίο ήθελε να στείλει στην Ουκρανία ένα φίλο σα και θα χρειαζόταν να πληρώσει πολύ ψηλά τέλη. Δυστυχώ τα πράγματα ακόμα δεν έχουν εξηγιανθεί απολύτω. Προφανώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα παρατυπιών. Και θα έλεγα στο φίλο σας όχι μόνο να γράψει σε εσά για το ζήτημα αυτό, αλλά να γύρει το ζήτημα αυτό με τι αρμόδιε αρχέ προκειμένου να γίνει προσφυγή ακόμα και στο δικαστήριο για τα ζητήματα αυτά, προκειμένου να φτάσει και στο δικαστήριο αυτή η περίπτωση δωροδοκία. Μόνο τότε θα δούμε απλά αποτελέσματα, για το πρόβλημα είναι ότι πολύ συχνά οι πολίτε απλώ παραπονούνται, αλλά δεν αναλώνουν τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να κάνουν καταγγελίε, προκειμένου να προχωρήσουν σε δικαστικέ προσφυγέ. Και αυτό ακριβώ θα πρέπει να κάναμε όλοι μα να αναλαμβάνουμε τέτοια δράση οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, οποιοδήποτε πόστο και αν έχουμε. Είτε εργαζόμαστε στο Κοινοβούλιο, είτε είμαστε πολιτικοί, είτε εκπροσωπούμε την κοινωνία των πολιτών. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ για τις πληροφορίες που μας δώσατε και για τη συζήτηση. Αυτό είναι το τελευταίο σημείο της διακοινοβουλευτικής ε, ε συνόδου. Αν θέλετε όμως να παραμείνετε, μπορούμε παρα, μπορείτε να παραμείνετε έχουμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κατάσταση στην Τουρκία. <coughs> Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το επόμενο σημείο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία. Γιατί τις τελευταίες μέρες έχουμε παρακολουθήσει με μεγάλη ανησυχία την κράτηση πολλών βουλευτών του κόμματος ΧΑΝΤΕΠΕ, του κόμματος Ελευθερίας των Λαών, μεταξύ των οποίων η Φιγγένη Στακ και ο Σελαχατίν Ντεμιρτάς. Το HDP είναι το τρίτο κοινοβουλευτικό κόμμα στην τουρκική βουλή και οι κρατήσεις των βουλευτών του είναι ένα μεγάλο πλήγμα στον πολιτικό πλουραλισμό στην Τουρκία. Εξάλλου, αυτό το μέτρο είναι κάτι που απομακρύνεται πολύ από τις αξίες και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Μούσνιξ, είναι μεγάλη χαρά το να μπορούμε να έχουμε την παρουσία σας σήμερα και βέβαια σας ε, καλέσαμε ευσπευσμένα ουσιαστικά και είχατε την ευγένεια να έρθετε ενώπιόν μας για να μας παρουσιάσετε τις απόψεις σας για τα πρόσφατα γεγονότα στην Τουρκία και ιδίως για την έκθεση για το που, αναφέρατε, που δημοσιεύσατε πρόσφατα για τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα των αποφάσεων που έλεγε η τουρκική κυβέρνηση με το κράτος έκτακτης ανάγκης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξοχότατοι κυρίε και κύριοι βουλευτέ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να έρθω ενώπιον σα. Είναι μια μεγάλη ικανοποίηση για μένα να ξέρω ότι ενδιαφέρεστε για αυτά που κάνουμε για την Τουρκία. Η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία είναι ένα θέμα μεγάλη ανησυχία για μένα και σε όλου μα στο Συμβουλίο τη Ευρώπη. Όταν βλέπω τον ευρύτερο, ευρύτερο χώρο του Συμβουλίου τη Ευρώπη, η Τουρκία είναι ένα σημείο καυτό σε ό,τι αφορά τα γεγονότα. Εγώ έχω πάει πέντε φορές στην Τουρκία τα τελευταία τέσσερα μισή χρόνια και είδαμε να υπάρχει μια πολύ σοβαρή επιδείνωση της τοπικής ειδικής κατάστασης. Έκανα μια επίσκεψη 9 ημερών τον Απρίλιο του 2016 και προετοίμαζα μια έκθεση για την Τουρκία όταν έγινε η απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο. Ξαναπήγα στα, στο τέλος Σεπτεμβρίου για μερικές μέρες και όπως είπε και ο πρόεδρος έχω δημοσιεύσει ένα μνημόνιο για τα μέτρα εκτακτής ανάγκης μετά από το πραξικόπημα. Το... Η προσπάθεια πραξικοπήματος ήταν βέβαια μια τραυματική εμπειρία και ήταν απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε και τις πηγές αυτού του πραξικοπήματος. Γι' αυτό το λόγο αυτό εγώ δεν διαμφισβητώ <clears throat> το γεγονός ότι η Τουρκία ε, κήρυξε κράτος έκτακτης ανάγκης και πήρε μια εξαίρεση από τους κανόνες της ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αλλά υπήρξε και μεγάλη ε, ασάφεια σε σχέση με αυτή την εξαίρεση. Δεν σημαίνει μια τέτοια εξαίρεση ότι πάβουν να ισχύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να ισχύει πάντα η αναλογικότητα στα μέτρα που λαμβάνονται και κάποια άρθρα τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν μπορούν να τύχουν εξαίρεση. Αυτή τη στιγμή έχει απόλυτη σχεδόν διακριτική ευχέρεια η εκτελεστική εξουσία στην Τουρκία και ο κίνδυνο αυθαίρετων ενεργειών είναι τεράστιο. Τα μέτρα αυτά έχουν επηρεάσει όχι μόνο το δημόσιο τομέα, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ προβληματικό. Τα μέτρα αυτά αποκλίνουν πολύ από τις φυσιολογικές διασφαλίσεις και υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες για το κράτος δικαίου εν γέννη, γιατί παραγωγικά το τεκμήριο αθωότητος, η, ο ατομικός χαρακτήρας της ε, ποινική ευθύνης η νομική ασφάλεια, η μη αναδρομικότητα του νόμου, η μη τιμωρία χωρίς ένδικη διαδικασία, η ισότητα όπλων σε μια δικαστική διαδικασία, όλα αυτά τα πράγματα έχουν σε μεγάλο βαθμό τεθεί ένα αμφιβόλο. Ακόμα και αν οι ευρείες εξουσίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση ήταν δικαιολογημένες αμέσως μετά την ε, απόπειρα πραξικοπήματος, αυτή η δικαιολογία μετά από την πάροδο του χρόνου είναι όλο και λιγότερο έγκυρο όσο απομακρυνόμαστε από τη χρονική στιγμή τη απόπειρα πραξικοπήματο. Τώρα έχουμε πάνω από 100.000 δημόσιου υπαλλήλου που έχουν απολυθεί, χιλιάδε ΜΚΟ και ε, ιδιωτικέ εταιρείε και οργανισμοί τύπου έχουν ε, πάψει να ισχύουν και αυτή η διαδικασία εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα. Αυτό το οποίο τονίζω στο μνημόνιο μου είναι ότι είναι απαραίτητο να αναστραφεί η λογική αυτή της έκτακτης ανάγκης και ο μαζικός τρόπος με τον οποίο έχουν δράσει η κυβέρνηση και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Μια άμεση ανησυχία ήταν οι σοβαρές καταγγελίες κακομεταχείρισης και βασανιστήριων μετά από την απόπειρα πραξικοπήματος. Αυτές οι καταγγελίες για κακομεταχείριση που φαίνεται ότι έχει λάβει χώρα ε, ήταν αποτέλεσμα της άρσης των βασικών διασφαλίσεων και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ένα αποφασιστικό σημείο όταν η υπηρεσία, η Επιτροπή μάλλον για την πρόληψη των βασανιστήριων στο Συμβούλιο της Ευρώπης θα διαβιβάσει την έκθεσή τους προς την τουρκική κυβέρνηση και τους έχουμε ζητήσει να το κάνουν αυτό το ταχύτερο δυνατόν για να υπάρξει σαφήνεια σε σχέση με το θέμα αυτό και για να μην υπάρχουν αμφιβολίες για το πόσο, κατά πόσο αυτές οι καταγγελίες ευσταθούν ή όχι. Τα κριτήρια για την ποινική ευθύνη σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ασαφέστατα. ΜΚΟ, ενώσεις πολιτών, τράπεζες, εταιρείε που συνδέονται με το κίνημα του Φετιουλαχ Γιουλέν είχαν λειτουργήσει με απόλυτα νόμιμο τρόπο μέχρι τις 15 Ιουλίου και δεν μπορείτε να τιμωρήσετε κάποιον γιατί αναδρομικά είχε κάποια σύνδεση με αυτή την οργάνωση όταν στις 15 Ιουλίου, μέχρι τις 15 Ιουλίου δεν ήταν έγκλημα το να συνδέεται κανείς με μια τέτοια οργάνωση σε ό,τι αφορά την αρχή της αναλογικότητας. Δεν μπορεί κανείς να εφαρμόσει την ίδια λογική στους δημοσίους υπαλλήλους, στα μέσα ενημέρωση, στις ΜΚΟ. Πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση έναντι του δημοσίου τομέα και έναντι του ιδιωτικού τομέα. Και μέσα στο δημόσιο τομέα δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε ένα δικαστή όπως ένα δημόσιο, με τον ίδιο τρόπο με ένα δημόσιο υπάλληλο σε ένα υπουργείο, γιατί δεν έχουν την δεν μπορούν να αποτελέσουν την ίδια απειλή προς το καθεστώς. Όλοι όμως αυτή τη στιγμή επηρεάζονται από αυτά τα μέτρα έκτακτης ανάγκης με ομοιόμορφο τρόπο. Οι ίδιες δραστικές κυρώσεις έχουν επιβληθεί, η ίδια λογική κολασμού έχει εφαρμοστεί, τα κριτήρια είναι ασαφή, υπάρχει έλλειψη παροχής αποδεικτικών στοιχείων που να είναι σαφή και αποφάσεις οι οποίες να είναι εξατομικευμένες. Θεωρώ ότι τα μέτρα αυτά τα οποία επηρεάζουν την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα είναι ιδιαίτερα προβληματικά, γιατί επηρεάζουν την ελευθερία του συνεταιρίζεστε και την ελευθερία της έκφρασης που είναι βασικές αρχές σε ένα οποιοδήποτε δημοκρατικό σύστημα. Η κατάσχεση στοιχείων ενεργητικού, η διάλυση οργανισμών χωρίς δικαστικές διαδικασίες, πιστεύω ότι είναι απόλυτα απαράδεκτη και απόλυτα δυσανάλογη. Μπορούν, εάν έχουν υποψίες, να αναστείλουν την ε, λειτουργία οποιοδήποτε οργανισμού και να παγώσουν τα στοιχεία του ενεργητικού αυτού του οργανισμού μέχρι την τελική δικαστική διαδικασία. Επίσης υπάρχουν προβλήματα με τα μέλη μιας οικο... της οικογένειας κάποιου υπόπτου. Πολλές φορές τα μέλη αυτά της οικογένειας κάποιου υπόπτου έχουν, έχουν αφαιρεθεί τα δικαστήριά του, τα διαβατήριά τους και έχουν παραβιαστεί άλλα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Αυτά είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Η δυνατότητα δικαστικής θεραπείας μέσα στην ε, Τουρκία είναι και αυτή ε, πάρα πολύ προβληματική. Υπήρξαν άτομα τα οποία απολύθηκαν γιατί βρισκόντουσαν σε ένα κατάλογο που είχε προσαρτηθεί ως παράτημα σε ένα νόμο και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν το δικαίωμα προσφυγής στο συνταγματικό δικαστήριο, δεν έχουν καμιά εθνική θεραπεία σε δικαστικό επίπεδο και δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνουν κάτι. Όλα αυτά οδήγησε σε μια πληθώρα περιπτώσεων ανθρώπων που προσπάθησαν να διαφυσβητήσουν αποφάσεις κυβερνήσεως εναντίον τους αλλά πολλές από αυτές τις περιπτώσεις έρχονται και στο ΕΔΑΔ στο Στρασβούργο. Υπάρχει μεγάλος αριθμός περιπτώσεων που έχουν υποβληθεί τις τελευταίες εβδομάδες και περιμένουμε να έρθουν και άλλες. Το να υπάρχει λοιπόν μια εσωτερική εθνική δυνατότητα θεραπεία προτού φτάσει κανεί στα διεθνή δικαστήρια, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία και για τη λειτουργία του συστήματο ω συνόλου το κατά πόσο τώρα η δικαστική εξουσία μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις ε, προσφυγές στην Τουρκία, αυτό είναι κάτι το οποίο υπόκειται σε σοβαρές αμφιβολίες. Όταν έχετε πάνω από 3.500 δικαστές και εισαγγελείς οι οποίοι έχουν απολυθεί η ανασταλή διαδικασία τους, η λειτουργία τους ή ακόμα είναι και υπόδικοι, είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η δικαστική εξουσία μπορεί να λειτουργήσει με αμερόληπτο τρόπο όταν ζήτησα από τι τουρκικέ αρχές πώ θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό, λένε «Α, θα στελεχώσουμε τις υπηρεσίες μας με νέους δικαστές και θα φέρουμε συνταξιούχου ε, δικαστές, θα του επαναφέρουμε στην υπηρεσία». Αυτό με κάνει πολύ σκεπτικιστή. Μετά από τη δημοσίευση του υπομνήματός μας, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω. Δύο νέα νομοθετήματα νομοθετικά διατάγματα, μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα, ένα από αυτά είχε ένα μεγάλο κατάλογο ατόμων τα, οι οποίοι θα απολυώσουν και ένα νέο διάταγμα περιορίζει ακόμα περισσότερο το δικαίωμα δικαστικής άμυνας των πολιτών μέχρι φτάνει να κρατούνται έξι μήνες στη φυλακή χωρίς πρόσβαση στην ε, φυλακή. Οι δύο συνδήμαρχοι του Διάρμπακερ έχουν κρατηθεί, που τους συνάντησα εγώ όταν ήμουν στην Τουρκία. Αυτό συνοδεύτηκε από ένα πάρα πολύ σημαντικό και προβληματικό ε, μέτρο που ήταν η αποκοπή 8 επαρχιών από το ίντερνετ σε 8 επαρχίες της Τουρκίας. Ελέγχθη ότι το ίντερνετ είχε πέσει σε αυτές τις περιοχές. Υπήρξε η επιδρομή κατά της Τζουμ Χουριέτ, της εφημερίδας αυτής πρόσφατα. Και εδώ είναι τόσο παράλογη Πόσο παράλογες και αυτές οι κατηγορίες που εκτοξεύστηκαν κατά της Τζουμ Χουριέτ, γιατί οι εκδότες της Τζουμχουριέτ κατηγορήθηκαν ότι ήταν και υπέρμαχοι του ΠΚΚ και γιουλενιστές. Αλλά αυτά είναι δύο πράγματα τα οποία είναι αλλοαποκλειόμενα. Παρ' όλα αυτά κατηγορούνται και για τα δύο. Και αυτό είναι για μένα σαφές δείγμα του γεγονότος ότι ο στόχος των μέτρων έκτακτης ανάγκης έχει τροποποιηθεί και έχει οδηγήσει σε καταχρήσεις. Έχουν κλείσει 15 ε, ραδιοσταθμοί και τηλεοπτικοί σταθμοί της ε, στο κουρδικού χαρακτήρα. Επίσης, η ασυλία των βουλευτών του Χαντεπέ για περιφρόνηση των δικαστηρίων έχει αρθεί η ασυλία τους με ένα πολύ προβληματικό τρόπο. Και εδώ η Επιτροπή Βενετίας, το συμβουλευτικό αυτό σώμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, θεώρησε ότι αυτό είναι κατάχρηση συνταγματικής διαδικασίας και δεν υπήρχε κανένας λόγος να μην αντιμετωπιστούν ατομικά οι περιπτώσει αυτών των ανθρώπων και όχι με συλλήβδιν τρόπο όπω έγινε στην πραγματικότητα. Ο διάλογο τώρα που έχω εγώ και το Συμβούλιο τη Ευρώπη με τι τουρκικέ αρχέ συνεχίζεται, αλλά αυτό ο διάλογο δεν έχει οδηγήσει σε κανένα αποτέλεσμα. Και είναι καιρό για την Τουρκία να δείξει κάποια δείγματα ανταπόκριση και σταματώ εδώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριο Καούσο, ο πρόεδρο, για τι πληροφορίε που μα δώσατε. Δίνω το λόγο στην κυρία Κάτι Πύρη που είναι συγγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Μουσνιξ διότι ήρθατε εδώ μετά από λίγη προειδοποίηση. Είπατε στο τέλος ότι τις δέκα τελευταίες μέρες, τις δέκα τελευταίες μέρες είδαμε την σύλληψη των δημάρχων του Διαρμπακύρ και είδαμε τόσους 142 δημοσιογράφοι το μεγαλύτερο αριθμό από όπου αλλού στον κόσμο που συνελήφθησαν και είδαμε και την σύλληψη 10 μελών ε, του τουρκικού κοινοβουλίου που εκπροσωπούν 5 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Δύο η ώρα το πρωί συνελήφθηκαν στο σπίτι τους και θεωρήθηκαν εγκληματίες ε, και φυλακίστηκαν. Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών βλέπουμε μια πτώση ε, στην Τουρκία, μια παρέκκληση από τις ευρωπαϊκές αξίες και η κατάσταση επιδεινώθηκε από το πραξικό σκόπιμα ε, και βλέπουμε πόσοι απολύθηκαν, πόσοι κρατούνται. Δεν, ε, τα με μίδια. Επίσης και βλέπουμε ότι η κουρδική μειονότητα δεν έχει έναν δημοκρατικό εκπρόσωπο, δημοκρατικούς εκπροσώπους που να έχουν μείνει ανέγγιχτοι. Βεβαίως το ΠΚΚ είναι στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Αλλά αν αφαιρέσετε από τους Κούρδους, τους δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους τους, θα μείνουν μόνο τα ριζοσπαστικά κινήματα των Κούρδων. Νομίζω ότι η Τουρκία κλείνει την πόρτα στην Ευρώπη. Η Τουρκία είναι εκείνη που κλείνει την πόρτα στην Ευρώπη και ακούμε ότι θα υπάρξει μια πρόταση από την τουρκική κυβέρνηση να προτείνει την επανεισαγωγή της θανατικής ποινής και αυτό κλείνει και την πόρτα στην Συμβούλιο της Ευρώπης και αυτό δεν μπορεί να παραμείνει χωρίς πολιτική απάντηση. Θα πρέπει, θα έχουμε και την συζήτηση αύριο στο Κοινοβούλιο όταν η Κομισιόν θα παρουσιάσει την ετήσια έκθεση της στο ερώτημα που σας θέτω. Σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας διότι είναι πάρα πολύ πολύτιμο για μας να έχουμε μια ανεξάρτητη γνώμη λεπτομερή, ενδελεχή, έναν συλλογισμό νομικό του τι συμβαίνει στη χώρα αυτή τι διαδικασία θα εισαχθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης εάν η Τουρκία την επόμενη εβδομάδα προτείνει νομοσχέδιο για την επανεισαγωγή της θανατικής ποινής. Τι αυτό θα σημάνει για την, το ότι είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης θα ανασταλεί το καθεστώς ε, του πλήρους μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης και όλες αυτές οι περιπτώσεις που λέτε ότι οι Τούρκοι πολίτες ακόμα και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τι θα συμβεί με αυτές τις περιπτώσεις στο χειρότερο σενάριο όπου ανασταλεί το καθεστώς μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αναφέρατε ε, την Επιτροπή Αποτροπής των Βασανιστήριων ε, και Κακομεταχείρισης. Ελπίζουμε ότι η Τουρκία θα δημοσιεύσει αυτή την έκθεση. Και μια τελευταία ερώτηση. Ξέρετε, τους τελευταίους μήνες συζητούμε συνέχεια για τον αντιτρομοκρατικό νόμο και επίσης ζητήσαμε κατευθυντήριες γραμμές από το Συμβούλιο της Ευρώπης προς την τουρκική κυβέρνηση. Ακόμα και αν γίνουν αλλαγές στην νομοθεσία ενώ υπάρχει η κατάκτασταση έκτακτης ανάγκης και βλέπουμε πώς υλοποιείται, θα αυτό ε, θα ε, απαντήσει στις ανησυχίες που έχουμε σχετικά με την ευρύτερη ερμηνεία αυτής της νομοθεσίας. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ μετά από τόσο σύντομη προειδοποίηση. Κυρία Σόμερ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω εξ ονόματος τη πολιτική μου ομάδα για την παρουσία σας, για το γεγονός ότι ήρθατε ενώπιον σας και σας ευχαριστώ επίσης και για τη σαφήνεια των λόγων σας βλέπουμε ότι έχουν αρθεί όλες οι διασφαλίσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλο και περισσότερο παρατείνεται και διευρύνεται. Ο Τούρκος πρόεδρος έχει επιτύχει αυτό το οποίο ήθελε ίσως, αλλά έχει καταστραφεί η δημοκρατία στην Τουρκία, δεν υπάρχει το κράτος δικαίου, έχει τεθεί εκτός παιδιάς τελείως το κράτος δικαίου ακόμα και δικαστές και εισαγγελείς βρίσκονται στη φυλακή, βρίσκει, δεν βρίσκει κανείς δικηγόρος πια. Και ακόμα και όταν ε, βρίσκει κάποιο ένα δικηγόρο, δεν τολμάει να εμφανιστεί ενώπιον των δικαστηρίων. Δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα να υπάρξουν πραγματικά νόμιμες διαδικασίε στα δικαστήρια. Δεν υπάρχουν νομικέ θεραπείε, όπω είπατε, και αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά όλου. Αλλά και πάλι θέλω να τονίσω ότι ήδη υπήρχε πριν από, την, ε, από, την, ε, ε, από το πραξικόπημα υπήρχε διαδικασία κατάσχεσης των στοιχείων ενεργητικού ορισμένων ιδιωτικών ομήλων και υπάρχει μια διαδικασία που ήδη έτρεχε πριν από το πραξικόπημα ενώπιον των δικαστηρίων. Υπάρχει λοιπόν και η περίπτωση αυτή για να επηρεαστούν τα μέλη της οικογένειας μιας ε, ενός ύποπτου. Δηλαδή κάποιος είναι υπόπτος και μετά η γυναίκα του ή τα παιδιά του τίθενται υπό παρακολούθηση ή ασκείται πίεση εναντίον τους, Υπάρχουν ε, επιχειρήσεις οι οποίες δημεύονται ουσιαστικά, περνάνε στο κράτος και Αναρωτιόμαστε σε τι μπορεί να οδηγήσει αυτό. Υπάρχουν καταστάσεις λοιπόν οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι αποδεικτές και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αναφερθήκατε και στο τεκμήριο αθωότητος. Εν τω μεταξύ λέγεται από πολλούς στην Ευρώπη ότι ναι μπορεί ο Γιούλεν να έχει κάνει αυτό το πραξικόπημα. Εγώ δεν έχω καμία συμπάθεια για αυτόν και την οργάνωσή του ούτε φυσικά και για το ΑΚΠ ή τον πρόεδρο του, αλλά, αλλά δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι το κίνημα του Γιούλεν ήταν αυτό το οποίο συμμετέσχε ή οργάνωσε το πραξικόπημα αυτό, την απόπειρα πραξικόπηματος και το να υπάρχει συλλήβδιν ε, υποψία όλων αυτών που συνδέονται με κάποιο τρόπο με το, κείμενο, κίνημα αυτό, αυτό μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει και στην Τουρκία να ισχύσει το τακμήριο ε, Αναφέρατε και ορισμένα άλλα σημεία. Έχουμε όλοι παρακολουθήσει τις εξελίξεις, κάτι το οποίο μας κάνει να ανησυχήσουμε πάρα πολύ και το είπε και η κυρία Πύρη προηγουμένως είναι οι υποψίες ότι γίνονται και πάλι ε, βασανιστήρια. Έχουμε ακούσει για κακοποίηση στις φυλακές, κακομεταχείριση και πρέπει να είναι πραγματικά ικτρές οι συνθήκες γιατί είναι απεριόριστες χιλιάδες ατόμων που έχουν συσσωρευτεί στις φυλακές. Έχουμε ακούσει για περιπτώσεις βασανιστήριων. Υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία φαίνεται ότι έχουν υποστεί πολλαπλές κακομεταχειρήσεις και είχαμε και την είδηση ότι ακόμα και οι ιατροδικαστές και ιατρικό προσωπικό έχει απολυθεί από τις θέσεις τους και αυτό μας κάνει να φοβόμαστε ότι είναι ακόμα ευρύτερο το πρόβλημα αυτό και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό το Συμβούλιο της Ευρώπης να αποκαλύψει όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα βασανιστήρια. Και γι' αυτό ε, συμμεριζόμαι αυτά που είπε και η συνάδελφή μου κάτι πήρη. Θα ήθελα και εγώ να θέσω το ερώτημα πώς θα αντιμετωπίσει το Συμβούλιο της Ευρώπης μια ενδεχόμενη ε, εφαρμογή της θανατικής ποινής και ίσως θα μπορούσε να μας δώσει και κάποια κατεύθυνση στο Συμβούλιο της Ευρώπης για το πώς πρέπει να δράσει η Ευρώπη. Παρακαλώ. Κύριος Μαυρίδης. <coughs> Uh, Έχω δύο ερωτήσεις βασικά. Δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαστική εξουσία στην Ταρκία. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Δεν υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακόμη περισσότερο. Χίλιοι, χιλιάδες απολύονται, συλλαμβάνονται, φυλακίζονται, βασανίζονται. Μια απλή ερώτηση. Όλα αυτά γίνονται και είναι ε, είναι αυτές προϋποθέσεις για μια δημοκρατία και ακόμα περισσότερο. Αν ε, δεν υπάρχουν, μπορούμε να πούμε ότι η Τουρκία επισήμως δεν είναι πλέον μια δημοκρατία. Αυτή είναι μια ερώτηση, διότι μπορούμε να μιλούμε συνέχεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε θεωρητικό πλαίσιο, αλλά τελικά ουσιαστικά όλα ε, καταλήγουν σε αυτή την απλή ερώτηση. Και η άλλη μου ερώτηση είναι η εξής. Συμφωνείτε μαζί μου ότι η ε, επιοίκεια που ακολουθήσατε τα τελευταία χρόνια έχει αποτύχει, ότι αυτή η γραμμή έχει αποτύχει και ότι πρέπει να βρείτε μια άλλη γραμμή απέναντι στην Τουρκία. Μήπως ε, θα πρέπει πρώτα να ζητήσουμε από την Τουρκία ε, να πληρεί όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Ο κύριος Χατζηγεωργίου έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω πως δεν χρειάζεται και εγώ να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για όλες τις πληροφορίες που μας έχει δώσει. Νομίζω ότι πρόσθεσαν στην εικόνα που μάλλον ήδη έχουμε όλοι και δεν θέλω ούτε εγώ να επαναλάβω όσα έχουν λεχθεί από εσά και από τους συναδέλφους που μίλησαν ως τώρα για τις φυλακίσεις, για τους βασανισμούς, για τις απολύσεις και πάνω απ' όλα την σύλληψη και τη φυλάκιση, αν είναι δυνατόν, του ηγέτη του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος της χώρας. Δύο μέρες μόλι, μόλις πριν το πραξικόπημα, σε μένα, εκπρόσωπος των δικαστών της χώρας, των δικηγόρων, με συγχωρείτε, της χώρας, μου είπε ότι ήδη έχουν στα χέρια τους κατάλογο με 2.000 δικαστές που θα απολύονται μέσα στις επόμενες μέρες. Και προηγήθηκε το πραξικόπημα, ήρθε το πραξικόπημα μάλλον, και μετά απελήθησαν αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω και ο κύριος Χάνο, επίτροπος διεύρυνσης, άφησε ένα αιωρούμενο <clears throat> πάνω σε αυτό το θέμα. Πώς ήταν δυνατόν να υπάρχει ήδη ο κατάλογος. Δεν θα πω εγώ ότι υπάρχουν θεωρίες συνωμοσία εδώ, αλλά ο κύριος Ερτογάν ο ίδιος έχει πει ότι το πραξικόπημα ήταν δώρο του Αλλάχ. Ένα ερώτημα μόνο μένει, γιατί οι επαναλήψεις και από εμάς και από εσάς η περιγραφή όλου του κακού που συμβαίνει στην Τουρκία, που εμείς ενδιαφερόμαστε για τον λαό της Τουρκίας, δεν, δεν προσθέτουν κάτι παραπάνω. Πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Και ένα λοιπόν είναι το ερώτημα. Τι σκέφτεστε να κάνετε. Και η αναφορά στη θανατική ποινή, εάν επέλθει λένε συνάδελφοι εδώ την επόμενη εβδομάδα, τότε θα πρέπει να πάρθουν τα πιο σκληρά μέτρα. Χωρίς καμιά αφιβολία Συμφωνώ 100%. Όμως εδώ σκοτώνονται άνθρωποι χωρίς, χωρίς δίκη. Χωρίς δίκη τους σκοτώνουν. Το ότι θα τους σκοτώνει και με δίκη ασφαλώς είναι ένα επιπρόσθετο ζήτημα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι δεν πρέπει να περιμένουμε και αυτό για να δείξουμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, το ερώτημα είναι τι θα κάνετε. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Λοκμπίλερ, δύο λεπτά παρακαλώ γιατί αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης για την έκθεση αυτή. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη για τη δουλειά που κάνουμε. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, όσον αφορά τα βασανιστήρια. Όταν μιλήσατε με τις τουρκικές αρχές, πώς σας εξήγησαν τα πράγματα, δηλαδή πώς δικαιολόγησαν τη χρήση της βίας και των βασανιστήριων. Όταν είχαμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης από την Τουρκία, απέφυγε να απαντήσει, είπα απλώς ότι η κυβέρνηση Ερντογάν θα πρέπει να την ευχαριστήσουμε γιατί έχει μία μηδενική ανοχή όσον αφορά τη βία. Πριν από κάποια χρόνια εγκρίθηκε αυτό. Επίσης μπορούμε να πούμε και η Επιτροπή Λειτουργία Αυτών με κ. Φαρογιάννης. Θέλω να ευχαριστήσω ε, τον Επίτροπο Μούσκινς ε, δεν έκρυψε τα λόγια του, ήταν πολύ σαφής στις περιγραφές του και δυστυχώς ε, συμπίπτουν και οι δικές μας απόψεις. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, Μικρή Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που είναι υποχρεωμένη ε, να συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, μία στην Τουρκία και μία στις Βρυξέλλες, παρά τις προσπάθειες που έχουμε κάνει και την σχεδόν ομόφωνη προσέγγιση που έχουν όλα τα μέλη όλων των κομμάτων που ανήκουν σε αυτή την Επιτροπή, δυσκολευόμαστε και παρά τους πολλούς συμβασμούς που κάναμε να βρούμε κοινό δρόμο συνεννόησης για να γίνει μετά από ένα χρόνο, ολόκληρο χρόνο αυτή η συνάντηση παρότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας έδωσε ειδική άδεια όχι μόνο να επισκεφτούμε την ε, Άγκυρα αλλά και να γίνει αυτή η Επιτροπή στην Άγκυρα παρότι ήταν η σειρά να γίνει στις Βρυξέλλες. Τώρα θέλω να θέσω και ένα ερώτημα. Πολύ σημαντικά όλα σε υπόθηκα και από τους συναδέλφους και από τον κύριο Επίτροπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, το κράτος δικαίου, τις διώξεις οι οποίοι υπάρχουν, τη θανατική ποινή. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση, η διάσταση της αμφισβήτησης ε, του, ε, του διεθνούς δικαίου, κυρίως με τη ρητορία του κυρίου Ερντογκάν, για την συνθήκη της Λοζάνης, μια διεθνή συνθήκη που καθορίζει τα σύνορα της Τουρκίας, το καθεστώς των στενών και την ανταλλαγή των πληθυσμών εκείνης της εποχής μεταξύ χωρών όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Τουρκία με ρητορία όπως τα σύνορα της καρδιάς μας, αναφορές στον όρκο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1920 ότι πρέπει να γίνουν δημοψηφίσματα για τις περιοχές που καταλάμβανε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή περιοχές από την Βιέννη μέχρι το Κυρκούκ, όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Αυτή η αυθαιρεσία η οποία υπάρχει στο εξωτερικό και περιγράφει και πάρα πολύ καλά από όλους τους ε, συναδέλφους να εξαχθεί και εκτός συνόρων. Και αυτό είναι το ερώτημά μου κατά πόσο ανησυχεί και το Συμβούλιο της Ευρώπης αυτή η προοπτική, αν συμφωνεί ο κ. Επίτροπος σε αυτή την ανάλυση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελένα Κύριε Βαλενθιάνο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Και εγώ δεν θέλω να επαναλάβω όλα αυτά που είπαν οι συναδελφοί μου, αλλά παραμένει η σημαντική αυτή η ερώτηση. Ποια είναι η άποψή σας ποια είναι η θέση, η θέση σας έναντι της δυνατότητας αναστολής της συμμετοχής της Τουρκίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης εάν εγκριθεί <clears throat> η επαναφορά της ε, θανατικής ποινής. Ποια είναι η θέση σας γενικά εναντί, εναντίον χωρών που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, το ερώτημα μου είναι το εξή. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό το οποίο θα έχει σημασία για τον Ερντογάν. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς το οποίο θα έχει κάποια επίπτωση στον ίδιο τον Ερντογάν. Εμείς ξέρουμε πάνω κάτω τι θέλουμε. Η θέση του Κοινοβουλίου μας είναι αρκετά συνενετική. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως που θα αγγίξει τον Ερδογάν χωρίς να πλήξει τους πολίτες της Τουρκίας και τους δημοκράτες στην Τουρκία. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, το οποίο πραγματικά θα ταρακουνήσει τον Ερδογάν χωρίς να θίξει τον λαό της Τουρκίας. Η κυρία Βεζιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και εγώ για τον απολογισμό αυτό που μας παρουσιάσατε όσον αφορά την κατάσταση στην Τουρκία. Συμφωνώ ότι η επιδείνωση ξεκίνησε πριν από την απόπειρα πραξικοπήματος, αλλά ότι η απόπειρα πραξικοπήματος αστικά βοήθησε να επιταχυνθεί αυτή η δικασία που είχε ήδη ξεκινήσει στο παρελθόν. Ανάμεσα σε αυτά που μας προκαλούν ανησυχία είναι ότι αυξάνεται ο εθνικισμός και κάθε φορά που οι Ευρωπαίοι λένε το παραμικρό, είτε στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρώπης, είτε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ε, υποστηρίζουμε αρκετά την Τουρκία. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο περνάει, ότι δεν υποστηρίζουμε αρκετά την Τουρκία απέναντι στο πραξικόπημα, ότι δεν υποστηρίζουμε εμεί Ευρωπαίοι την Τουρκία όσον αφορά την τρομοκρατία και ότι προσπαθούμε να την εκβιάσουμε. Αυτό είναι δυστυχώ το μήνυμα το οποίο περνάει τελικά στην Τουρκία. Εσεί στο Συμβούλιο τη Ευρώπη έχετε την ίδια εντύπωση όσον αφορά τη συμμετοχή δηλαδή της Τουρκίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ποια είναι η εντύπωση που έχετε εσείς επ' αυτού. Επίσης, ποια είναι η δική σας άποψη όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιδράει η Τουρκία στις ίδιες αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχω την εντύπωση ότι δεν αντιδρά πολύ καλά. Και τέλος, κάτι ακόμα σημαντικό όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τον ορισμό της τρομοκρατίας. είμαστε πολλοί εδώ πέρα, αλλά και ως το Συμβούλιο της Ευρώπης, που αναφερθήκαμε στην υφιστάμενη νομοθεσία που είχαμε στην Τουρκία, την αντιτομοκρατική και τη νέα μορφή που παίρνει, η νέα νομοθεσία με τη νέα πρόταση που έχει γίνει. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό και επίση αν μπορείτε να μα απαντήσετε για την επαναφορά τη ποινή, πιθανή επαναφορά τη αντική ποινή. Ο κύριο Μποργέζιο, θα ήθελα και εγώ να σε ευχαριστήσω για την σημαντική αυτή παρουσίαση. Δύο πολύ σύντομε ερωτήσει. Πρώτον, Η γενικότερη τάση είναι αυτή η επιδείνωση της κατάστασης, μια τάση θρησκευτικού ισλαμικού εξτρεμισμού στην Τουρκία. Και βλέπουμε ότι επομένως και στην Τουρκία θα μπορούσαν να ξεκινήσουν και περαιτέρω διώξεις των χριστιανών. Γιατί ξέρετε ότι επιλείται και η ίδια η θρησκεία εκεί υπάρχουν κάποια ανεσχετικά στοιχεία συγκεκριμένα τα οποία να έχετε εντοπίσει εσείς και αν ναι, τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε την ανεξιθρησκεία με συγχωρείτε στην Τουρκία και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των χριστιανών και των άλλων θρησκευμάτων. Πιστεύετε επίσης ότι υπάρχουν όλο και περισσότεροι κίνδυνοι σε μια χώρα για τους Ευρω... που δεν σέβεται πλέον το κράτος δικαίου για τους ίδιους τους Ευρωπαίους πολίτες, για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εκεί ή για τους ανθρώπους που μεταβαίνουν στην Τουρκία ακόμα και προσωρινά για επαγγελματικού λόγους. Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να, να προλάβουμε κάποιους περιορισμούς της ελευθερίας των ίδιων των Ευρωπαίων πολιτών αυτή τη φορά που ενδεχομένως να πηγαίνουν στην Τουρκία προκειμένου να εκφράσουν μια κάποια έμπρακτη ή πολιτική αλληλεγγύη προς αυτούς που διώκονται. Και ο κύριος Μπρόκ για να κλείσει η συζήτηση. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω δύο φράσεις για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές ότι οι τωρινές εξελίξεις μέσα στην Τουρκία έχουν οδηγήσει στο να απομακρυνθεί περισσότερο η Τουρκία από τη δυνατότητα να γίνει κάποτε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ μακρύτερα τώρα από μια ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι πριν από δύο ή πέντε ή δέκα χρόνια. Λόγω των εξελίξεων που έλαβαν χώρα στην Τουρκία. Είτε τότε, ήδη τότε το 2004 είχα επικρίνει την <clears throat> δυνατότητα ένταξης της Τουρκίας γιατί Είχα πει ότι τότε δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν εφικτό με τις τότε συνθήκες. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπεροχή της πολιτικής έναντι του, των στρατιωτικών <clears throat> και η κατάσταση τώρα αυτά. Έχουμε μια κατάσταση που κανείς δεν είναι ανεξάρτητος από κανένα, ανάλογα εκτός από τον πρόεδρο παρά μόνο ο πρόεδρος. Είναι ακριβώς μια αναστροφή της κατάστασης. Είχα την εντύπωση ότι, ότι οι μεταρρυθμίσεις θα οδηγούσαν σε ένα σύστημα το οποίο θα έφερνε πιο κοντά την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι έχει καταργηθεί το κεμαλιστικό σύστημα για να, δημιουργήσει, να θέση του ένα άλλο σύστημα το οποίο είναι ακόμα λιγότερο συμβατό με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν ε, εφαρμοστεί η θανατική ποινή στην Τουρκία, αυτός είναι ένας απε, απερίφραστος λόγος για την λήξη των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία για την ένταξη. Πρέπει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση όχι να αναστείλουμε, αλλά να περατώσουμε τις διαπραγματεύσεις. Δεν έχουμε άλλο εργαλείο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν μπορούμε όταν τίθενται τόσοι άνθρωποι στη φυλακή και παραβιάζεται κάθε μορφή ελευθερίας έκφρασης να ανοίγουμε κεφάλαια με την Τουρκία. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, δεν μπορούμε να αφήσουμε να γίνονται εκτελέσεις στην Τουρκία και εξάλλου μέσα στην εντολή του Συμβουλίου προς την Κομισιόν λέει ότι μπορεί να είναι το τέλος της διαδικασίας η ένταξη της Τουρκίας, αλλά εάν προκύψουν δυσκολίες στο δρόμο, σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να επιστήσουμε απλώς την καλύτερη δυνατή σχέση με την Τουρκία. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε κατά πόσο είναι αξιόπιστο να έχουμε μια διαφορετική άποψη από αυτό που ήταν η εντολή της Τουρκίας. Η Τουρκία βέβαια το να χαθεί από την Ευρώπη και να περάσει σε ένα Ισλαμιστικό στρατόπεδο δεν είναι κάτι που είναι προς το συμφέρον μας. Ε, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της Συρίας, το θέμα των ε, προσφύγων θέλουμε να συνεργαστούμε και με την Τουρκία και με την Αίγυπτο και με την Τινησία. Δεν είναι κάτι που είναι προς το συμφέρον μας να χάσουμε αυτή τη δυνατότητα συνεργασίας. Πρέπει λοιπόν να να μην έχουμε <clears throat> μια λύση η οποία θα επιτρέψει στα τρία εκατομμύρια Σύρων που βρίσκονται στην Τουρκία να φέρουν αυτή το βάρος αυτής της απόφασης και να μην έχουν την σωστή α, από την Τουρκία. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν του θέματος της ε, ε, ένταξης να λάβει υπόψη και όλες τις άλλες πτυχές της σχέση της με την Τουρκία και όχι να τα βάλει όλα στο ίδιο καλάθι. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μούσνιξ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις Μερικές είναι κάπως πολιτική, πολιτικές και είναι εκτός της δικής μου εντολής που αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά θα αναφερθώ σε αυτές τις ερωτήσεις που αφορούν ιδιαίτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η θανατική ποινή μας ανισχύει. Δεν μπορεί κανείς να είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και να έχει θανατική ποινή. Μπορεί κανείς βεβαίω να κάνει πολλά πράγματα και να μείνει μέλος, όπως το απέδειξε το πρόσφατο παρελθόν, αλλά όχι θανατική ποινή. Νομίζω ότι αυτό θα προκαλέσει συζήτηση ε, στα πολιτικά όργανα, στην Επιτροπή ε, Υπουργών, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Δεν θα είναι μια συζήτηση στην οποία εγώ θα συμμετέχω. Ε, θα είναι πολιτική συζήτηση και για μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι ένα πράγμα που κανείς δεν μπορεί να κάνει και να παραμείνει στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Όχι το μόνο, αλλά ένα από τα σημαντικά που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το καθεστώς του μέλους θα είναι ε, κατάφορο διάβημα κατά ε, μιας αρχής συμπεφωνημένης από όλους. Όλα τα άλλα μπορεί κανείς να τα παρακάμψει, αλλά όχι αυτό να τα αλλοιώσει. Όσον αφορά τα βασανιστήρια, υπήρχαν πολλοί ισχυρισμοί βασανιστήριων, κυρίως αμέσως μετά το πραξικόπημα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επαληθευθούν, να εξυμβρωθούν το ότι δεν έχουμε ένα μηχανισμό εθνικό προληπτικό μέσα στην Τουρκία, αλλά νομίζω ότι με το υλικό που έχει η κυβέρνηση για το πραξικόπημα υπονομεύει την περίπτωση της κυβέρνησης. Παραδείγματος χάρη είπα, ε, το πρακτορείο Ανατολού που είχε πολλές φωτογραφίες που τις έδωσε ε, ε, τις φωτογραφίες αυτές αεροπορικές εταιρείες σχετικά με το πραξικόπημα και σε μια φωτογραφία βλέπετε κάτι που είναι σαφώς κακομεταχείριση. Βλέπετε στρατιωτικούς οι οποίοι είναι κάτω στο έδαφος γυμνοί. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και αυτό είναι στο υλικό της κυβέρνησης που διανέμεται. Αυτό ήταν ε, μια μεγάλη success story. Η, Τουρκία πρόδευσε πάρα πολύ στην καταπολέμηση των βασανιστήριων με τη συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ήταν ένα σημείο που είπα στις ε, τουρκικές αρχές, μην χάσετε αυτό το υπέρ, αυτή την επιτυχημένη ιστορία της συνεργασίας μας. Μην θυσιάστε αυτό το επίτευγμα να λάβετε σοβαρά υπόψη τα πράγματα. Ε, βεβαίως διαψεύδουν τους ισχυρισμούς και, ε, και θα τους είπα ε, ότι αυτά τα μέτρα, το να περιορίζετε την πρόσβαση σε δίκη χώρο ε, το να αλλάζετε τον τρόπο που στις φυλακές γίνονται οι ιατρικές εξετάσεις, το να κρατάτε τα άτομα απομονωμένα χωρίς καμία επικοινωνία. Αυτές είναι περιπτώσεις κακής μεταχείρισης. ότι υπάρχει μαζική, μαζικά βασανιστήρια, δεν μπορώ αυτό εγώ να το ισχυριστώ. Ε, θα δούμε την έκθεση της Επιτροπής Πρόληψης Βασανιστήριων τι θα συμβεί εάν ε, γίνει κάτι με το καθεστώς μέλους της Τουρκίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι, οι περιπτώσεις θα εξεταστούν και θα, ε, θα τις παρακολουθεί η Επιτροπή Υπουργών. Ακόμα και αν αυτές ε, οι περιπτώσεις αυτές ε, τις, οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο θα μελετηθούν για να δούμε τι θα γίνει με το καθεστώς του μέλους. Η κοινωνία των πολιτών τώρα. Πώς θα στείλουμε ένα μήνυμα στην η πολιτική ηγεσία να υποστηρίξει την κοινωνία των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών αισθάνεται παραμελημένη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματά τους ξεχάστηκαν από τους φίλους της Ευρώπης, κυρίως στην νότια ανατολική περιοχή και οι άνθρωποι εκεί αισθάνονται ότι ε, δεν, ε, δεν ασχοληθήκαμε αρκετά με, την, ε, με, τις, με τα blackout, με την απαγόρευση κυκλοφορίας κλπ. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών στις σχέσεις με τις αρχές. Αυτό που προσπάθησα να πω στις αρχές και επανειλημμένα τους είπα, χωρίς πολλή επιτυχία μέχρι τώρα. Έχουν ε, μεγάλους ε, πόρους, έχουν μικιό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουν ενώσεις επαγγελματικές δικηγόρων, γιατρών που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, πανεπιστημιακούς και όλοι αυτοί συνεργάζονται. Και η κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν τους, θεω, δεν τους δίνει την αξία που έχουν. Θα πρέπει και αυτοί να μιλήσουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα θέματα σχετικά με τα σύνορα είναι πολιτικό θέμα. Διώξεις των χριστιανών δεν είδα εκθέσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Με διώξεις μεγάλης κλίμακας δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, αλλά δεν πέσυρε κανείς την προσοχή μου πάνω σε αυτό. Η κίνδυνη για τους Ευρωπαίους πολίτες τη μέρα τον Απρίλιο που έφυγα από τον Διαρμπακύρ έγινε μια επίθεση τρομοκρατική, μια επίθεση ό,τι πιστέψει κανείς για τον Γκιουλέν είναι, υπάρχουν τρομοκράτες οι οποίοι δρούν στην Τουρκία του ΠΚΚ, της ΔΑΕΣ και άλλοι τρομοκράτες που είναι πραγματικός κίνδυνος και απειλή. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τις πράξεις της κυβέρνησης στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και αυτό είναι το θέμα σε ένα μνημόνιο που θα αναφερθεί το Δεκέμβριο σχετικά με την αντιτρομοκρατία στην νότιο-ανατολική Τουρκία. Θα δούμε την νομιμότητα των μέτρων, την αναλογικότητα, την νομολογία σχετικά με την αντιμορισία των υπηρεσιών ασφαλείας στην έλλειψη των ερευνών, των ανακρίσεων, παραλληλισμοί με προηγούμενες περιπτώσεις, με ομάδες περιπτώσεων, με την ατιμορρησία, με τους ισχυρισμούς. Το επόμενο βήμα από μένα είναι αυτό το μνημόνιο ε, για την αντιτρομοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην νοτιοανατολική Τουρκία. Έκθεση θα δημοσιευθεί ε, το Δεκέμβριο. Ε, τον Ιανουάριο ελπίζω ένα άλλο κείμενο για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και δεν νομίζω ότι αλλάζοντας την, την διατύπωση του νόμου κατά της ε, τρομοκρατίας αλλάζει την κατάσταση. Το θέμα είναι πώς η δικαιοσύνη εφαρμόζει την νομοθεσία. Πολύ συχνά βλέπουμε τα απλά σημεία αναφοράς με τα οποία μπορούμε να κρίνουμε την πρόοδο ή όχι. Αλλά το θέμα είναι πιο περίπλοκο πώς η εισαγγελία και η δικαιοσύνη ασχολείται με τις περιπτώσεις αυτές και θα, αν ενδιαφέρεστε για την μοίρα των ηγετών της ΧΑΝΤΕΠΕ υπάρχει μια καλή περίπτωση από την αρχή ε, της ε, περίπτωσης του DDP που ήταν ε, προκάτοχος του ΧΑΝΤΕΠΕ και η Τουρκία έχασε την υπόθεση αυτή στο δικαστήριο και εκεί βασικά είχαμε την ευρύτερη αντίληψη της αντιτρομοκρατίας κατά της απαγόρευσης ενός κόμματος και είναι το θέμα το οποίο εσείς αναφέρατε, ότι δηλαδή ότι οι ειρηνικές επιλύσεις των διενέξεων και ο προσδιορισμός της κουρδικής ταυτότητας είναι μορφές νόμιμες ελεύθερης έκρευσης. Και φημώνοντας αυτές τις ε, φωνές αφήνεται το πεδίο ελεύθερο για αυτούς που κρατούν τα όπλα και αυτή είναι επικίνδυνη πορεία, επικίνδυνος ο δρόμος και βλέπουμε ότι τα μέλη του ΧΑΝΤΕΠΕ έχουν, ε, υπήρξαν θύματα όπως και ακτιβιστές, ε, όπως και δημοσιογράφοι είναι ε, μια καμπή αρνητική των γεγονότων. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ασχολείται εντατικά με την Τουρκία, συνεργάζεται. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα έρθει την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο θα έχω μαζί του μια συνάντηση και ελπίζω ότι η έκθεση της Επιτροπής κατά της, των βασανιστήριων θα δημοσιευθεί σύντομα. Έχουμε βουλευτές στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση που κάνουν παρόμοια εργασία και βεβαίως το δικαστήριο συνεχίζει τη δουλειά του. Χαίρομαι που βρήκατε το κείμενό μου χρήσιμο. Είναι σημαντικό να μιλάμε με μία φωνή από την ίδια βάση και ελπίζω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε την Τουρκία να αλλάξει πορεία, να αποσύρει αυτά τα μέτρα και να ασχοληθεί με τις σοβαρές ανησυχίες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπάρχουν σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε και κλείνουμε αυτό το σημείο. Meine Damen und Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συναδελφοί, η πρότασή μου είναι να αναβάλουμε την εξέταση της έκθεσης για τον ΟΗΕ, να έρθουμε στην έκθεση για τη Μογγολία, που έχει, πιστεύω, προτεραιότητα. Κύριε Σόλτς, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι η Μογγολία είναι στις ε, χώρες του κόσμου που από τη δεκαετία 1990 έχουν περάσει μια βαθιά πολιτική και κοινωνική μεταρρύθμιση έχει προχωρήσει σε μια νέα οργάνωση της οικονομίας της με την κρατική κατα... καθοδήγηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να αναπτύξει μια σωστή, ένα σωστό πλαίσιο συνεργασίας μαζί με τη Μογγολία. Το 2013 οδήγησε αυτή η διαδικασία σε μια συμφωνία συνεργασίας και τώρα έχουμε μια ευρύτερη συμφωνία συνεργασίας και εταιρική σχέσης. Η διαδικασία κύρωσης αυτής της διαδικασίας μεταξύ των κρατών μελών πλησιάζει το τέλος, την περάτωσή της είναι τρία κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακόμα δεν έχουν κυρώσει αυτή τη συμφωνία. Πρέπει ακόμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει τη συνέγκρισή του για να ανοίξει το δρόμο για μια πιο στενή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μογγολίας. Έχουμε μια καλή παράδοση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να συνοδεύουμε αυτές τις διαδικασίες με ένα ψήφισμα. Και έχοντας αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, έχω την εντύπωση ότι αυτό το ψήσιμο μπορεί να είναι και μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε με διαφοροποιημένο τρόπο την εξέλιξη στην Μογγολία και να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η προοπτική συνεργασίας με την ε, Μογγολία και το σχέδιο μου λοιπόν ψηφίσματος είναι στη διάθεσή σας. Ακολουθούμε βέβαια τους κανόνες η οποία είναι πολύ αυστηρή σε σχέση με το μήκος αυτού του ψηφίσματος. Δεν ξεπερνάει λοιπόν τα όρια αυτά το ψήφισμά μας και προσπαθεί να διορθώσει το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε <clears throat> ασχοληθεί αρκετά με την Μογγολία. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να θεσπίσουμε και να εδραιώσουμε σχέσεις με τη Μογγολία που θα οδηγήσουν σε πραγματική συνεργασία. Η Μογγολία, και το λέω αυτό, σαφώς θα πρέπει να αποδεχθεί τους κανόνες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι απαραίτητο να ακολουθήσει το ευρωπαϊκό παράδειγμα σε ό,τι αφορά την δημοκρατική πορεία και εξέλιξή της από την ε, δεκαετία του 1990 για πρώτη φορά το πολιτικό σύστημα της Μογγολίας χαρακτηρίζεται από μια ειρηνική εναλλαγή στην ε, ε, εξουσία. Μπορεί κάποια από αυτά τα στοιχεία να είναι μονάχα τυπικά, αλλά παρόλα αυτά η εκλογική διαδικασία έχει οδηγήσει σε κάποιες πραγματικές αλλαγές. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι <clears throat> μια πλήρως ανεπτυγμένη χώρα σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Επομένως, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ακόμα ότι θα συμμορφωθεί η Μογγολία με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και με προδιαγραφές σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να ακυρώσει τα αντίστοιχα νομικά εργαλεία. Και μας ενδιαφέρει βέβαια και ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστούν αυτές οι προδιαγραφές στην ε, πράξη. Μας ενδιαφέρει επίσης να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα των ε, <clears throat> δημοσίων αρχών και επίσης θέλουμε να ενισχύσουμε και τη δυνατότητα καλύτερης ε, ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών. Και επίσης να ενισχύσουμε την διαίρεση των εξουσιών θα πρέπει να ξεπεραστεί η ασάφεια των κανόνων που έχουν να κάνουν με τα κόμματα και τις δραστηριότητές τους. Επίσης, το σχέδιο νόμου που έχει να κάνει με τις κοινοβουλευτικές εκλογές θα πρέπει να επανεξεταστεί και ενδεχομένω η Μογγολία να προχωρήσει σε τροποποίηση σε σχέση με αυτό το νομοθέτημα. Είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί και ο ποινικό κώδικας και μια σειρά μέτρων όπως η θανατική ποινή η οποία θα πρέπει να καταργηθεί. Είναι θέματα τα οποία είναι πάντα προσφολή στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο. Μετά από την έκθεση της Transparency International για την διαφθορά, η Μογγολία δεν είναι πια στις τελευταίες σειρές των κρατών, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η έκταση της διαφορά στη Μογγολία είναι κάτι το οποίο αφορά και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και των πόρων του υπεδάφους της Μογγολίας και εξάλλου η κοινωνική και η οικονομική πολιτική που έχει ακολουθήσει η Μογγολία έχει οδηγήσει σε σε μια πολιτική για τους φυσικούς πόρους που οδήγησε σε, μια μεγάλη, σε ένα μεγάλο χάσμα για, μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού βρίσκεται κάτω από το κατόφλι της Ένδειας και η οικονομική ανάπτυξη δεν έχει καταφέρει να μειώσει αυτή την ψαλίδα. Ένα μικρό μέρος μονάχα του πληθυσμού έχει την εξουσία πάνω στους φυσικούς πόρους και τον πλούτο της χώρας. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να οδηγήσει σε ένα κράτος δικαίου και σταθερότητα. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει στο ότι η ανεργία <clears throat> έχει μειωθεί στην χώρα αυτή και ένα πολύ μεγάλο μέρος του ενεργού πληθυσμού μπορεί να έχει μια απασχόληση, περίπου 85%. Έχει μειωθεί, η, έχει αυξηθεί μάλλον η, το εξωτερικό χρέος σε 83% και τα αποθεματικά βρίσκονται τώρα σε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Για επειδή δεν έχει τα απαραίτητα αποθεματικά για να καλύψει τις ανάγκες της το 2017, η Μογγολία έχει απευθυνθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσει η κυβέρνηση της ε, Μογγολίας πώς θα εξασφαλίσει την ε, εξυγίανση αυτού του χρέους, γιατί αυτό κινδυνεύει να οδηγήσει σε κοινωνικές εκρήξεις και να τροφοδοτήσει μεταναστευτικά κύματα από τη Μογγολία σε άλλες χώρες και επίσης μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ιδιαίτερα επιβάλλησης του περιβάλλοντος. Επομένως, μια αναλλακτική αντιμετώπιση θα πρέπει να επιλεγεί από την <clears throat> κυβέρνηση της Μογγολίας, η οποία μπορεί μονάχα με την μεγαλύτερη ενσωμάτωσή της σε περιφερειακά σχήματα ολοκλήρωσης να βελτιώσει την κατάστασή της. Στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει μια, ένας μετασχηματισμός της ε, οικονομίας της ε, Μογγολίας και επίσης να αναπτυχθεί με τους άμεσους γείτονές της μια διαδικασία συνεργασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια καλύτερη κατεύθυνση της χώρας αυτής, ώστε να διαχειριστεί καλύτερα την εξωτερική της πολιτική έναντι της ε, Ρωσίας και της Κίνας και να έχει μια πιο ανεξάρτητη πολιτική από ό,τι είχε επιτευχθεί μέχρι τώρα. Φαίνεται ότι η πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει αντιμετωπίσει αυτή την ε, πραγματικότητα. Πολλά κράτη μέλη όπως η Γερμανία έχουν κατευθύνει την πολιτική τους μόνο υπό το πρίσμα των οικονομικών σχέσεων. Επομένως δεν εκπλήσει κανένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι μετά από τη μονογραφή της ε, συμφωνίας ε, εταιρική σχέσης μέχρι την τελική της κύρωση έχουν περάσει σχεδόν 6 χρόνια. Και θέλω να τονίσω προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι εμείς θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτήν την συμφωνία γιατί θα βοηθήσει τη Μογγολία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά που ανέφερα και η εφαρμογή αυτή της συμφωνίας θα πρέπει να συνοδεύεται από την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αρρωγεί στην Μογγολία να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα τα οποία ανέφερα. Και επομένως θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία να υπάρξει μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση στην περιοχή και επίσης θα πρέπει να δράσουμε με πραγματιστικό τρόπο για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που είχε η μέχρι τώρα πολιτική στην Μογγολία. Και τέλος, θα πρέπει να αποφασίσουμε να έχουμε στην Ουλάν Βατόρ μια ευρωπαϊκή <clears throat> αντιπροσωπεία και να ενισχύσουμε και τον τη συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου της Μογγολίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ προσβλέπω λοιπόν στη συζήτηση η οποία θα μπορέσει να λάβει χώρα εδώ και την περαιτέρω συνεργασία που ελπίζω θα είναι καρποφόρα. Dankeschön. Σας ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος, ο κύριος Κέλεμ. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Να εκφράσω την υποστήριξή μου για το κείμενο του συναδέλφου Χέλμουντ Σόλ. Συμφωνώ με την προσέγγισή του. Είναι εκτενές πλήρες το κείμενο και εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λεκού Κόμματος μπορώ να πω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε την προσέγγισή του. Διότι η Μογγολία φαίνεται για πάρα πολλούς μια πολύ απομακρυσμένη, κατοικημένη χώρα. Στην πραγματικότητα όμως έχει έναν κέριο στρατηγικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην περιοχή. Αποτελεί γέφυρα μεταξύ των μεγάλων κρατών της Ασίας, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Και σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο αυτή η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μογγολίας είναι καθοριστικής σημασίας και πραγματικά μπορεί να δεσμεύσει περισσότερο την Μογγολία στην τήρηση του κράτους δικαίου. Ήδη έχει δεσμευθεί κατά θετικό τρόπο η Μογγολία στην εδραίωση της δημοκρατίας και όπως είπε και ο συνάδελφος Σόλς πριν από λίγο, ήδη η Μογγολία στην Κεντρική Ασία θεωρείται ένα πρότυπο πλέον δημοκρατικού μετασχηματισμού. Ξέρουμε ότι είναι μια περιοχή με πάρα πολλά προβλήματα. Η Μογγολία επίσης δραματίζει έναν ρόλο οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην όλη περιοχή. Και αυτό χάρη στο ουδέτερο καθεστώς, χάρη στον διάλογο που υπάρχει στα πλαίσια του Λαν Μπατόρ και όσον αφορά τώρα την οικονομία της χώρας. Η Μογγολία αυτή τη στιγμή βρίσκεται ανάμεσα σε διαφορετικά οικονομικά σχέδια όπως ο δρόμος του μεταξιού της Κίνας, βρίσκεται κοντά στους ενεργειακούς διάβλους της Ρωσίας είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μογγολίας να λειτουργήσει ομαλά και να μην παρεποδιστεί αν η Μογγολία τελικά μπήκε στην ε, Ευρωσιατική Ένωση. Ε, αυτό είναι ένα ακόμα μήνυμα το οποίο θα πρέπει να στείλουμε μέσα από την έκθεσή μας. Συνεπώς, η Μογγολία χρειάζεται μια θετική δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια εμβαθυμένη, ενισχυμένη συνεργασία. Από πλευρά μου θα πρότεινα κάποιες ε, περαιτέρω ιδέες. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να έχουμε μια ειδική συνεργασία με τη Μογγολία όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ας μην ξεχνάμε επίσης την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την ελευθερία έκφρασης, ζητήματα πολύ σημαντικά για την εδραίωση της δημοκρατίας. Η εμπορία ανθρώπων είναι μια ακόμα ανησυχία που εξακολουθούμε να έχουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση, μολονότι έχουν ληφθεί μέτρα και μια συγκεκριμένη νομοθεσία κατά της εμπορίας ανθρώπων πριν από τέσσερα χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο στο πρόβλημα αυτό. Και τέλος, θα σας πρότεινα να παράσχουμε επιπλέον χρηματοδοτική βοήθεια στη Μογγολία για την επένδυση σε νέες τεχνολογίες, τεχνολογίες ψηφιοποίησης. Αυτό με τη σειρά του θα μπορούσε να συμβάλλει στην κάλυψη των αναπτυξιακού χάσματος που εντοπίζουμε αυτή τη στιγμή στη Μογγολία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ο συνάδελφός μου δεν είναι εδώ και θα διαβάσω αυτό το σημείωμα γι' αυτόν. Θα ήθελα να με συγχωρέσετε που δεν είμαι παρόν σήμερα, αλλά υποχρεώσεις με ανάγκασαν να γυρίσω στην Ιταλία νωρίτερα. Ε, χαίρομαι που παρακολουθώ τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας με τη Μογγελία εκ μέρους της Ομάδας Σοσιαλιστών Δημοκρατικών και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Σόλτς για το σχέδιο έκθεσης του οποίου συμμερίζομαι το θετικό τόνο το Κοινοβούλιο ε, θα πρέπει να δώσει την συνένεσή του ε, σε αυτήν την ε, συμφωνία που υπογράφτηκε από την Επιτροπή το 2013 που ακολουθήθηκε με επικυρώσεις βραδίες από τα κράτη-μέλα που δεν ολοκληρώθηκαν. Πρέπει να επιταχύνουμε την διαδικασία. Περιμέναμε πάρα πολύ καιρό για να προοδεύσουμε στην εταιρική μας σχέση με αυτό το στρατηγικό εταίρο. Είναι δημοκρατική χώρα ε, ε, μια χώρα που στρέφεται προς την Ευρώπη λόγω των κοινών μας αξιών, της ειρηνικής φύσης της χώρας και της ε, τάσης για πολυμερή συνεργασία. Είναι στρατηγικός εταίρος για την Ευρώπη και θα πρέπει να γίνει αυτό όπως γίνεται και με την πολιτική με τρίτες χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα. Ε, λόγω της αναβολής ε, προς όφελος χωρών όπως η Ιαπωνία και η Καναδά που αυξάνουν την ε, παρουσία τους εδώ, δημιουργήθηκε ένα κλίμα δυσπιστίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε τέτοιες εταιρικές σχέσεις με πολλές χώρες της Κεντρικής Ασίας, ενώ εδώ τώρα ε, προσπαθούμε στο Λαμπατάρ να ολοκληρώσουμε τη σχέση και η αποστολή Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται ακόμα από αυτήν ε, του Μπέιτζιν. Θα πρέπει να, να επιταχύνουμε τη συνεργασία με την ε, Μογγολία τώρα που έχει μια οικονομική κρίση, υπάρχουν και προκλήσεις επειδή, μετά την πτώση των φυσικών πόρων. Μπορούμε να δούμε μερική, μερικά σημάδια ανάκαμψης με τη νέα κυβέρνηση που προσπαθεί να αναστρέψει την κατάσταση. Επίσης υπάρχει μεγάλη ανάγκη για διαφοροποίηση της οικονομίας. Πρέπει να υποστηρίξετε τη Μογγολία σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό Νομίζουμε ότι θα πρέπει αυτή η εταιρική σχέση συνεργασίας να αποτελέσει ένα νέο βήμα στην εταιρική μας σχέση. Ο Charles Τάνοκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι είναι καλά εξισορροπημένη η έκθεση του κυρίου Σόλτς. Εγώ αγωνίστηκα με τη δική μου ομάδα στο, στη συνέλευση των Πρόεδρων για να καλέσουμε στο Στρασβούργο τον Πρόεδρο της Μογγολίας για να λάβει το λόγο και είχαμε μια πολύ καλή ευκαιρία μαζί με τον κύριο Μπρόκ να με τον κύριο Ελμπεκτότς δεν, δεν μπορώ να προφέρω το όνομά του σε θαυμάσια αγγλικά και εγώ εντυπωσιάστηκα από το όραμα που έχει για τη χώρα του που γιορτάζει τα 20 χρόνια δημοκρατίας. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ σε αυτή την εξωτική και μακρινή χώρα αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι μια χώρα που χρειάζεται τη βοήθειά μας, είναι πλουραλιστική, έχει τεράστιους φυσικούς πόρους που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, ένα μικρό πληθυσμό μονάχα, θέλει, σύμφωνα με τον πρόεδρό της, η χώρα αυτή να ακολουθήσει μια πολυπολική πολιτική και γνωρίζει την, ε, τις, ε, ε, τάσεις των δύο μεγάλων γειτόνων του που θέλουν να παίξουν ένα ηγεμονικό ρόλο στην ε, Μογγολία. Είναι λοιπόν μια χώρα που θέλει να έχει καλύτερες σχέσεις και με τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το κόμμα το ΕΣΥΑ δεν έχει κανένα πρόβλημα να υποστηρίξει την εταιρική και ε, σχέσεις συνεργασίας με τη Μογγολία και να αναπτύξει καλύτερες σχέσεις. Ευχαριστώ. Για την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η κυρία Γιακόφσκα έχει το λόγο. Παρακαλώ. χωρίς μικρόφωνο. Εκπροσωπώ. Ονομάζω Μαϊκόφσκα και αντιπροσωπεύω την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για τις σχέσεις με την Ασία, τη Μογγολία. Σας ευχαριστώ για τα γενικά σας λόγια υποστήριξης είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας ότι μπορούμε να βασιστούμε πάνω στην υποστήριξη στην βοήθεια σας. Από ό,τι καταλαβαίνω, ένας από του τομείς που δεν αφέρθηκε άμεσα, αλλά που θα έπρεπε να αναπτυχθεί και να αντικατοπτρίζεται περισσότερο σε μελλοντική συνεργασία στη σχέση μας μεταξύ των Κοινοβουλίων Μογγολίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα θέμα που ήδη αρχίσαμε, στο οποίο αρχίσαμε ήδη η προπαρασκευαστική εργασία, το διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι που βρίσκεται σε τροχιά και ελπίζουμε ότι του χρόνου θα αρχίσουμε αυτόν τον νέο μηχανισμό συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι κλείνει το θέμα της Μογγολίας. 11 Νοεμβρίου το μεσημέρι προθεσμία για τις τροπολογίες. 5 Δεκεμβρίου θα ψηφίσουμε. Και κατά πασχεδότητα θα πάμε στην Ολομέλεια τον Φεβρουάριο. Τελευταίο σημείο. Με την παράκληση να είμαστε σύντομοι, γιατί και εγώ έχω μια περαιτέρω συνεδρία που θα πρέπει να προεδρεύσω στις 6.30. Είναι η επίσκεψη στην Γεωργία στις 30 ε, Οκτωβρίου για το δεύτερο γύρο των κοινοβουλευτικών εκλογών είχαμε εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων με επικεφαλής την Άννα Γκόμες ε, μέσα στα πλαίσια της αποστολής της ΟΑΣΕ και με την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΟΑΣΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και το ΝΑΤΟ. Ιάννα, Να ευχαριστήσω καταρχήν τα μέλη της ομάδας μας και, το, και τη γραμματεία που βοήθησαν να δημιουργηθεί ένα καλό ε, κλίμα με την αποστολή της, ε, του, της ΟΑΣΕ και τις άλλες κοινοβουλευτικές συνελεύσεις στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Είχαμε ήδη συσσωρεύσει αρκετή γνώση για τις διαδικασίες της εκλογικές. Όλα πήγανε καλά στα εκλογικά τμήματα. Έξω από τα εκλογικά τμήματα μερικές φορές σε κάποια σημεία ήταν κάπως τεταμένη κατάσταση, επειδή υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι θέλαν ενδεχομένως να εκφοβήσουν τους ε, ψηφοφόρους. Υπήρξαν και άλλες ε, άλλα παράπονα για προσπάθειες ε, εκφοβισμού, αλλά αυτά δεν μπορέσαμε να τα επαληθεύσουμε. Είδαμε ακριβώς το ίδιο που είδαμε και την πρώτη φορά. Υπήρξε πολλές φορές ε, συνοστισμός στα εκλογικά τμήματα που δεν φαίνεται να είναι ένα τυχαίο φαινόμενο. <clears throat> πολλές φορές αυτό θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα παρέμβασης στην εκλογική διαδικασία. Οι εκλογικές επιτροπές ήταν κυρίως γυναίκες, έκαναν μια εξαιρετική εργασία. Αυτό το οποίο επίσης σε αυτά τα Επισόδια τα οποία αναφέραμε και τονίσαμε ότι όλα αυτά δεν ήταν τέτοια μορφή ώστε να πούμε ότι η έκφραση της λαϊκής θέλησης αυτών που πήγαν να ψηφίσουν ότι δεν αλλοιώθηκε. Κάποιες πολιτικές σκέψεις τώρα που μπορώ να εκθέσω. Δεν χρειάζεται τώρα να παραγνωρίσουμε αυτά τα θέματα το θετικό είναι ότι τα πράγματα πήγαν γενικά ειρηνικά και ομαλά, πέραν κάποιων επεισοδίων, ιδίως στην προεκλογική εκστατεία. Υπήρξαν ε, οι ανάγκες επανάληψης των εκλογών σε ορισμένε περιοχές. Παρ' όλα αυτά τα αποτελέσματα έγιναν αποδεκτά, παρά τις επικρίσεις οι οποίες διατυπώθηκαν από εκπροσώπους κομμάτων που δεν είχαν τη δυνατότητα κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης μετά από, τα, από τις εκλογές. Η μείωση όμως του, του φάσματος του πολιτικού που εκφράζεται, που συμμετέχει στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας δεν είναι ένα καλό φαινόμενο. Ενώ, εντάξει, υπάρχουν και χώρες που έχουν μονάχα δύο κόμματα στο Κοινοβούλιο, εν πάση περιπτώσει συρρυκνώθηκε το πολιτικό φάσμα το οποίο εκπροσωπείται στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας και κάτι άλλο το οποίο ήταν ενοχλητικό ίσως για ορισμένους είναι ότι η τρίτη πολιτική δύναμη στο Κοινοβούλιο δεν αποκρύπτει τους δεσμούς της με τη Ρωσία και, τον, και το αντιδραστικό της θεματολόγιο. Ένα άλλο στοιχείο αυτών των εκλογών ήταν και το γεγονός ότι υπήρξε μια πλειοψηφία η οποία επιτεύχθη από το κόμμα της, ε, το οποίο ε, είναι στην εξουσία και όλα αυτά εναποθέτουν μια μεγάλη ευθύνη στο κόμμα το οποίο έχει την εξουσία ώστε να εξασφαλίσει ότι αυτή η κοινοβουλευτική ε, πλειοψηφία δεν θα οδηγήσει σε αντίπεινα κατά των αντιπάλων της και για την περαιτέρω συρρήκνωση του πολιτικού τοπίου. Αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ ε, σημαντικές ε, για τη δημοκρατία, αλλά η δημοκρατία πρέπει να ασκείται και ενδιάμεσα, ανάμεσα στις εκλογές. Θα πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, ε, ελευθερία έκφρασης και αυτό δεν ε, συμβαίνει πάντα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μέσα στα πλαίσια των εκλογικών διαδικασιών. Και πρέπει να πω κλείνοντας ότι είμαστε σε μια χώρα όπου η παρακολούθηση των εκλογών και η διάδρασή μας με τους ε, τοπικούς παράγοντες ήταν πάρα πολύ σημαντική. Γιατί όλοι τους χαιρέτησαν το ρόλο μας και την παρουσία μας και επομένως δεν θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε σχέση με τη δυνατότητα να είμαστε ειλικρινείς εναντί των φίλων μας της Γεωργίας και να τους πείσουμε να, αποδεθούν σε ένα πραγματικό πολιτικό διάλογο ο οποίος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εξαρτίας ήταν κάπως περιορισμένος και είναι απαραίτητο να εργαστούμε με έναν τρόπο συνεργατικό, να εργαστούμε με έναν συνεργατικό τρόπο στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας και κατά την άποψή μου είναι μια πρόταση που σας υποβάλλω, θα πρέπει να ενισχύσουμε την συνεργασία μας με το Κοινοβούλιο της Γεωργίας και τους εταίρους μας, δίνοντας έτσι συνέχεια στην έκθεση αυτή που θα εκθέσουμε, θα εκδώσουμε για την, τις εκλογές, ξεπερνώντας και τα θέματα των εκλογών και αυτό περιλαμβάνει όλα αυτά τα θέματα τα οποία ανέφερα προηγουμένως όπως είναι η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις που <clears throat> μας έδωσε μεγάλη ικανοποίηση το να είμαστε μέλη μιας αντιπροσωπείας όπου οι συνομιλητές μας και από το κόμμα της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης γενικά αναγνώρισαν το ρόλο μας και ήταν έτοιμοι να ακούσουν τις απόψεις μας <clears throat> και τη δική μας ανάγνωση των προβλημάτων και των ευκαιριών που ανοίγονται μπροστά μας. Ήταν χρήσιμη αυτή η αλληλεπίδραση. Ευχαριστώ. Και εγώ επειδή ήμουν στον πρώτο γύρο μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, κυρίως την Αννα Γκόμες, επικεφαλής της ομάδας και τα μέλη της γραμματείας που ήταν πολύ επαγγελματίες και βοήθησαν πολύ σε αυτή την επίσκεψη. Ήταν αρκετά μια πλήρης εμπειρία. Η Γεωργία έχει προτεραιότητα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Ευρωπαϊκών κρατών δικαίως και θα ήθελα να αναγνωρίσω την αξία της εργασίας μας, των εκθέσεών μας ε, και βεβαίως όπως παρουσίασε τα πράγματα η αναγκόμες στο τέλος της αποστολής μας μαζί με τις άλλες οργανώσεις που συμμετείχαν και θα έλεγα ότι η έκθεση αυτή είχε πραγματική αξία και ίσως από τις πιο λεπτομερείς ε, που υπέδειξε πάρα πολλές προβληματικές απόψεις ε, αυτών των εκλογών. Υποστηρίζω πλήρως την προκαταρκτική δήλωση όπως παρουσιάστηκε στο, στην Τυφλίδα και θα ήθελα να τονίσω την δύσκολη εκστρατεία, προεκλογική εκστρατεία. Υπήρξαν πάρα πολλοί ε, τομείς εκφοβισμού περιπτώσεις εμφοβισμού, ε, συμπεριφορές εχθρικές και η χρήση διοικητικών μέσων. Βεβαίως θα θέλαμε, δε, κανείς δεν ήθελε να αμφισβητήσει ε, τα αποτελέσματα των ε, εκλογών, αρχίσει συζητήσεις με τα μέλη της αντιπολίτευσης οι οποίοι ε, υποστηρίζουν ε, την αξία της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης, αλλά θα ήθελα να κάνω έκκληση ε, στην, στο κυβερνών κόμμα, διότι είδα πολλούς νέους φιλοδυτικούς, νέους με πολύ καλή εκπαίδευση που απογοητεύτηκαν από αυτές τις εκλογές και είναι από τους μεγαλύτερους θησαυρού μιας χώρας σχετικά μικρής. Θα πρέπει να ενθαρρυθούν, να ληφθούν υπόψη και να έχουν τα δικά τους μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνήντησα νέους δικηγόρους που εκπροσωπούν τον σύλλογό τους και πάρα πολλοί θεωρούν ότι αυτές οι εκλογές αντίθετα με αυτό που είδαμε ε, στην ημέρα των εκλογών ε, και στα ε, ήταν λίγα και θα ήθελα να κάνω έκκληση στην κυβέρνηση της Γεωργίας να, ότι πρέπει να τους διαβεβαιώσει, να τους δώσει προοπτική στο μέλλον κάτι το πρόσθετο, υπάρχει ακόμα ένα κενό τον εκλογικό νόμο. Πάρα πολλοί συνομιλητές, ακόμη και εμπειρογνώμονες του ΑΣΕ, παρατηρητές, μίλησαν για ακατάλληλες νομικές διατάξεις περιγράφοντας τον δεύτερο γύρο της διαδικασίας. Ήτανε αυτονόητο ότι ε, στο τελευταίο στάδιο το προεκλογικό πριν από το δεύτερο γύρο σε αυτήν την περίοδο οι πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές ε, από την Κεντρική ε, Εκλογική Επιτροπή ήταν αναγκαίες και ήταν το μόνο φως για πολλούς προέδρους επιτροπών και ήταν ανάγκη να αλλάξει ο εκλογικό νόμο. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιο άλλο να θέλει να λάβει το λόγο. Μπορούμε να κλείσουμε και αυτό το σημείο και θα ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι συμμετέσχαν σε αυτή την άσκηση. Θα συνεχίσουμε την παρακολούθηση το θέμα των διαφόρων. Δεν υπάρχει τίποτα από μένα. Η επόμενη συνεδρίασή μας στις 14 Νοεμβρίου στις 3 η ώρα το απόγευμα. Καλό βράδυ.